Philippe. Mr. De Backer. Okay. Um, well, well... Λοιπόν, καλώ ήλθατε στη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα, Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, παρά το γεγονό ότι δεν έχουμε <clears throat> όλου του σκιώδει εδώ. Ελπίζω ότι θα έρθουν και θα προσφέρουν και αυτή τη συνεισφορά τους πριν από το τέλος της συζήτησης. Είμαστε στο σημείο 6, η βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις μικρό επιχειρήσεις και θα δώσω το λόγο στον Φιλίπ Ντεμπάκερ που είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ξέρετε η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό επηρεάζει τους επιχειρηματίες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αρχή του χρόνου η Κομισιόν παρουσίασε ένα σχέδιο βελτίωσης χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με καλύτερη πρόσβαση, περιλαμβάνει ενδιαφέρουσε πληροφορίες και επιλογές <clears throat> και διάφορες προτινόμενε λύσεις. Συζητήσαμε αυτό το σχέδιο δράση και την τωρινή κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με πολλούς εμπλεκομένους, επιχειρηματίες των μικρομεσαίων και είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε σε επαφή με τα τεκτενόμενα επίσης και με οργανώσεις των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ. Θεωρούμε ότι είναι θετικό το κείμενο της Κομισιόν, θα προτιμούσαμε περισσότερη άμεση δράση και πιο συγκεκριμένα και απτά μέτρα. Μετά από την κρίση, η Κομισιόν δεν έχει, κατά την άποψή μα, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση τη κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδίως για την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να παρατηρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να έρθουν κατεπηγόντω και να παρουσιάσουν συγκεκριμένε προτάσει. Δεν χρειαζόμαστε νέε προτάσει, χρειάζεται μια βελτιοποίηση, βελτιστοποίηση <clears throat> πρακτικών σε άλλα κράτη-μέλη πολλέ φορέ και αυτό μπορεί να είναι επαρκέ. Γι' αυτό οι δικέ μου προτάσει δεν είναι επαναστατικού χαρακτήρα. <clears throat> Χρειάζονται και από τι δύο πλευρέ βελτιώσει και από την πλευρά των επιχειρηματιών και από την πλευρά της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ζητάμε να υπάρχει πιο επαγγελματικός χαρακτήρας για τους επιχειρηματίες. Πολλές φορές δεν έχουν βασικές γνώσεις της λογιστικής, της ε, διαδικασίας χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη συζήτηση μεταξύ επιχειρηματιών και τραπεζικών φορέων. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των χρηματοδοτών, δεν υπάρχει κατανόηση των ειδικών συνθηκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλές φορές δεν υπάρχει και διαφάνεια για το λόγο για τον οποίο απορρίπτονται αιτήσει χρηματοδότησή τους. Πιο αργά. Για την ίδια τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Πολλά μπορούν να λεχθούν. το σχέδιο δράσης, το οποίο έχει προτείνει η Κομισιόν, ορθά δίνει έμφαση στο κεφάλαιο κινδύνου. <clears throat> Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση εύκολα προσβάσιμη σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το κλειδί για τη βελτίωση χρηματοδότησης είναι η πολυπικιλία. Αναφέρω το λεγόμενο crowdfunding, την χρηματοδότηση από πάρα πολλές πηγές, το οποίο μπορεί να είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να εξασφαλίσει το κεφάλαιο σερμαγιάς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αδρανούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλύτερη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι φορεί, λοιπόν, οργανώσει και κυβερνήσει κατανοούν τη σημασία τη καλή πρόσβαση σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στι επιχειρήσει αυτέ και σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν Συμπράξει δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για καλύτερη χρηματοδότηση. Προσβλέπω σε συνεργασία με όλους σα, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε συγκεκριμένε προτάσει και να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα προς τα εμπρός στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Καλώς. Ο κύριο Ντόρφμαν. Ähm, σας ευχαριστώ. Θέλω ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του και για πάρα πολλά σημεία υπάρχει απόλυτη σύμπνοια με τον εισηγητή και δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε. Είναι ζωτική σημασία στο να μπορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, κάτι που είναι δύσκολο ακόμα και σε φυσιολογικές οικονομικές συγκυρίες. Είναι γεγονός ότι πολλοί επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν αρκετή γνώση και κατάρτιση για τα θέματα αυτά Επομένως, είναι δύσκολο να ε, εποφελθούν της αγοράς πίστοσης, αλλά πολλές φορές έχουν και δυσκολία να παρουσιάσουν εγγυήσει για τη δανειοδότηση και είναι σε υποδέστερη θέση από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά επειδή βρισκόμαστε τώρα σε μια ιδιαίτερη οικονομική κρίση, είναι ακόμα μεγαλύτερες οι απαιτήσει από την πλευρά των τραπεζών για χρηματοδότηση από την άλλη μεριά οι εγγύσεις που μπορούν να δώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν συρρυκνωθεί και σε πάρα πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια οικονομική συγκυρία η οποία ε, διατρέχεται από απεσιοδοξία σε σχέση με το μέλλον. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα κάτι το οποίο ξεφεύγει και από τα στενά όρια αυτής της έκθεσης. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τι είναι πιο ενδιαφέρον για μια τράπεζα να δώσει πιστώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια αυτά για επενδύσεις σε χρηματιστηριακές πράξεις. Μια τράπεζα θα κάνει αυτό το οποίο είναι το πιο κερδοφόρο. Και προς το παρόν φαίνεται ότι είναι οι επενδύσεις στις χρηματαγορές, δυστυχώς. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον και προσοδοφόρο για τις ε, τράπεζες αυτό το οποίο όμως θα έπρεπε να γίνει για να χρηματοδοτήσουν καλύτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι να κάνουν πιο ελκυστικέ τι πιστώσει προ τι ΜΜΕ. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Για τι ε, συγκεκριμένε τώρα περιπτώσεις που αναφέρει ο εισηγητής θα ήθελα να σταθώ μονάχα σε τρία σημεία. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι σαφές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μεθοριακές ε, περιοχές είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της ψαλίδας επιτοκίων. Κάτι το οποίο οδηγεί σε πολλά προβλήματα και μειονεκτήματα ανταγωνισμού για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκεί όπου το, η διαφορά των επιτοκίων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Κάτι ακόμα το οποίο μου φαίνεται πολύ σημαντικό μέσα στην πρόταση της Κομισιόν είναι το ερώτημα σε ποιο βαθμό εμείς είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και σε συγκεκριμένα βήματα σε σχέση με, ένα, με συστήματα συλλογικών εγγύησεων κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν κράτη-μέλη όπου υπάρχουν συστήματα πίστοσης με συνεταιρισμούς ε, πίστης κατά κάποιο τρόπο, με συλλογικές εγγυήσεις από ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που με τον τρόπο αυτό μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό θα ήταν χρήσιμο να σκεφτούμε κατά πόσο θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε ένα τέτοιο σύστημα στην Ευρωπαϊκή, στη σύνολη Ευρωπαϊκή Ένωση και με την αρρωγή της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και εν κατακλείδη μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της πολιτικής πληροφόρησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολλές φορές δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν και έχουν άγνοια και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σαν στόχο να ευνοήσουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε λίγο καλύτερα για το πώς θα μπορέσουμε και μαζί με τα πιστοτικά ιδρύματα που ασχολούνται με τον τομέα αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε <clears throat> μια καλύτερη προσφορά πληροφοριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να ευνοήσουμε την πρόσβασή τους στην αγορά πίστης. Και κατά τα άλλα συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία έχει αναφέρει ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια εξαιρετική έκθεση. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τα θέματα τα οποία παρουσίασε. Αυτό που είναι σαφές από το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει εμείς να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα θέματα τα οποία έχουν δημιουργήσει οι τελευταίες αποφάσεις στα πλαίσια της νέας αρχιτεκτονικής της μικρομεσαίας. Ίσως θα πρέπει να θυμίσουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την βασική αρχή που λέγει ότι τα μικρά αντιμετωπίζονται πρώτα. Πρέπει δηλαδή να λάβει περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα των μικρομεσαίων στις αρχές του σχεδιασμού της πολιτικής της έτσι ώστε η πολιτική αυτή να είναι φιλική στους χρήστες. Και σε σχετικά με τα μακροοικονομικά μέτρα αυτά θα πρέπει να τεθούν στην πρώτη γραμμή. Για το περιεχόμενο έχω καταθέσει ορισμένες τροπολογίες Υπάρχουν διαφορε... Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης για τους διαφορετικούς τύπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής ότι είναι δύσκολο αν όχι ε, επικίνδυνο να αντιμετωπίζονται οι μικρομεσαίες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν μπορούμε να έχουμε τη λογική του ένα νούμερο κάνει για όλους ε, συνολικά αποδεκτή. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να προσπαθήσουμε να πιέσουμε ε, και την πρωτοβουλία μικροπιστώσεων. 100 εκατομμύρια προβλέπονται στα πλαίσια του προϋπολογισμού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, μέχρι και το 2014. Από το 2014 μέχρι το 2017 ξέρουμε ότι προετοιμάζει μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει προβλέψει ένα δις για την κάλυψη προγραμμάτων όπως του προγράμματος καινοτομίας και κοινωνικής αλλαγής και το 20% των ποσών αυτών θα προέλθει από μακροχρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτά τα σημεία συμπίπτουν, αν θέλετε, με τα θέματα των venture capital. Ε, σχετικά με τα ταμεία αυτά θα ήθελα να πω επίσης ότι θα πρέπει να, συνδεθούν και με τον κοινωνικό τομέα δραστηριοποίησης της επιχειρηματικότητας, βασικός στόχος της, ε, ε, του προγράμματος για την Ευρώπη 2020 είναι μια βασική προτεραιότητα και αυτήν επιδιώκω με τις τροπολογίες μου. Και τέλος, ε, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και το πόσο μπορεί να επηρεάσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιφερειακή πολιτική. Όλα είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο γιατί τα επόμενα 7 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εντείνει την χρήση αυτών των νέων καινοτόμων μέσων ιδιαίτερα στα πλαίσια της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτά. Um, Philippe. Yes, it's your Philippe, η σειρά σου. Πάνω στην ώρα. Να απαντήσεις, να απαντήσεις ε, σε όλα. Ποιος, ο Ντεκ πρώτα. Ευχαριστώ. Εγώ μιλάω εκ μέρους του κύριου Καμάλ, ο οποίος ε, επισκέπτεται, τώρα βρίσκεται μάλλον στη διάσκεψη του κόμματός του στο Μπέρμιγχαμ. Ναι, το κόμμα συνεδριάζει στο Μπέρμιγχαμ και ποιος ξέρει τι θα συζητήσουν τότε για τον κοινοτικό προπολογισμό εκεί. Κάποια μέρα ελπίζω ένα βέτο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο κύριος Καμάλ ευχαριστεί τον ε, εισηγητή και την Επιτροπή για την πρότασή της, αλλά τονίζει και ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συγχρόνως αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη. Ε, χαίρεται που βλέπει ότι ο εισηγητή υπογραμμίζει την ιδιαίτερη φύση της αγοράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει βέβαια ένας ενιαίος ορισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βασίζεται ανατομέα για την ε, ανακεφαλοποίηση στην αγορά, για, ανάλογα με τους απασχολούμενους κτλ. Γι' αυτό και πιστεύει ότι προσπαθώντας να ε, καταλήξουμε σε μια λύση που να ταιριάζει σε όλους, κάνουμε λάθο. Γιατί κάθε μικρομεσαία επιχείρηση αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα. Είτε πρόκειται για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είτε πρόκειται για την απασχόληση, να βρει κατάλληλο προσωπικό κτλ. Επίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα από τα πιο αποτελεσματικά επίπεδα για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει να κάνει με το εθνικό επίπεδο. Είδαμε στο Λονδίνο μεγάλη επιτυχία όπου εκατοντάδες επιχειρήσεις κίνησης κατάφεραν πριν ε, από λίγα χρόνια να ξεκινήσουν και να έχουν μεγάλη επιτυχία μέσα στις ειδικέ ε, συνθήκες του Λονδίνου. Είναι πράγματα μερικές φορές για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα, οπότε μην το παρακάνουμε στις φιλοδοξίες μας. Παρ' όλα αυτά βέβαια υπάρχουν μερικά χρήσιμα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα να ολοκληρώσουμε ρυθμίσει από τις οποίες να μπορούν να αποφεληθούν οι startup επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως ε, είναι οι ρυθμίσει για τα κοινοπραξίες ε, κλπ. Ο κύριος Καμάλ θέλει να συνεργαστεί με τον εισηγητή, με τον κύριο Ντεμπάκερ, για αυτό το θέμα, παρόλο που ε, πιστεύει ότι δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα να τροποποιηθούν. Αυτά. Κατά τα άλλα μένει στον εισηγητή. Ωραία. Φιλίπ. Ευχαριστώ Σαρών. Ζητώ συγγνώμη. Γιατί ο, ο Φιλίπ Λαμπέ δεν ήταν γέρος, Γι' αυτό θα προσπαθήσω να σε εξηγήσω τι πρόκειται. Ο συμπατριώτης μου <clears throat> και συνονόματός μου Φίλιπ έχει κάνει πολύ καλή εργασία. Θέλω να τον ε, συγχαρώ και να τον ευχαριστήσω. Τέσσερις παρατηρήσεις σε σημεία που μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Πρώτον, τα κίνητρα για την καινοτομία. Συμφωνώ μαζί του ότι πρέπει να έχουμε κάποιο παράγοντα έλξης κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ο αριθμό των μέτρων και των κανονισμών που αποφασίζουμε Παραδείγματο χάρη, παίρνουμε το, την αυξανόμενη αποδοτικότητα στη χρήση ενέργεια ή τη μείωση του διοξιδίου του άνθρωπο. Αυτοί είναι παράγοντε οι οποίοι έχουν το χαρακτήρα όθηση. Αλλά δεν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πιέσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προχωρήσουν στη γενοτομία. Πρέπει να τις ε, ενθαρρύνουμε, αλλά να έχουμε και δεσμευτικά μέτρα. Χρειαζόμαστε σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο ομάδων μέτρων να θέλουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή γενικότερα επιχειρήσει να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα. Ένα καλό παράδειγμα είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Θυμηθείτε ότι επιχειρήσει να αποφεύγουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες στα δεσμευτικά μέτρα, καθυστερεί η καινοτομία. Και τελικά δεχτήκαν ότι εφόσον δεν μπορούν σε επίπεδο αυτορύθμισης να πετύχουν στόχους, πρέπει να δεχτούν τις <clears throat> επιβαλλόμενες ρυθμίσεις. Επίσης, λες Φίλιππ ότι οι ψηλότεροι ε, λόγοι κεφαλαίου, ε, ποσοστά κεφαλαίου θα οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά έχουμε πολλές τράπεζες στην Ευρώπη ε, και στο Βέλγιο ιδίως η Τρίοδος, η Φανμπρέντα, συνεχίζουν να ε, δανείζουν επιχειρήσεις ενώ έχουν φτάσει το επίπεδο της, που απαιτεί η Βασιλεία 3. Ένα βασικό θέμα είναι το θέμα της ταχύτητα. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε από τα κεφαλουχικά επίπεδα που έχουμε τώρα σε αυτά που πιστεύουμε ότι θέλουμε να φτάσουμε, τότε ουσιαστικά αναγκάζουμε τις τράπεζες να μειώσουν τους ισολογισμούς τους και όχι να βελτιώσουν την κεφαλουχική τους επάρκεια. Είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσουμε στα, στους στόχους μας. Ε, παίζει ρόλο για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, θα δούμε τον κύριο Ντράγκη σε λίγο. Και υπάρχει το θέμα της αιρεσιμότητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναφέρει πολύ συχνά. Ο κύριος ε, Ντράγκη. <clears throat> Χρησιμοποιούμε ε, υποστήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όταν χρησιμοποιούμε μη πρότυπα εργαλεία θα πρέπει να υπάρχει κάποια αρεσιμότητα η οποία συνοδεύει αυτές τις ενέργειες. Και τέλος, ακόμα και αν δεν είναι αρμοδιότητα πλήρως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει η Κομισιόν και να μας στείλει και κάποιο σχετικό έγγραφο για τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την παρότρινση για χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά προγράμματα στην, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια καλύτερα από τα άλλα. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε αν η Κομισιόν χωρίς να δαπανίσει εκατομμύρια ευρώ για κάτι τέτοιο, να μας φέρει μια έκθεση και να εξηγήσει ποιο κάνει τι και ποιε είναι κατά την άποψή του οι καλύτερε πρακτικέ. Σταματάω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο Ζων, Ζων Πολ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τι προτάσει του και τα σχόλιά του. Κάποιες απλές και απλή λογική παρατηρήσεις. Το θέμα της χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχω αρχίσει και γερνάω, το ακούω πάντα, όπου και αν είμαι παρά τις περίπλοκες σκέψεις των ειδικών δεν έχουμε λύσει τίποτα. Δεύτερον, ποιος μπορεί να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες. Τρεις πηγές. Πρώτον, ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ο οποίος θα συνεισφέρει με τα δικά του μέσα, περιορισμένα συνήθως. Δεύτερον, οι τράπεζες, για τις οποίες πολλά λέμε. Και τρίτον, οι επενδυτές. Όμως σήμερα, οι τρεις αυτές πηγές έχουν στερέψει, σχεδόν στερέψει οι τράπεζες για τους λόγους που είπαμε, ενώ όταν βλέπουμε βέβαια τους αριθμούς ε, από κοντά ότι ε, τα δάνεια προς την οικονομία είναι πιο σημαντικά από τις καταθέσεις που παίρνουν οι τράπεζες, τουλάχιστον για τις γαλλικές τράπεζες. Και ο επενδυτής είναι ένα είδος στην ανεπαρκία. Για τα risk capital Νομίζω ότι σε τρία χρόνια δεν θα έχουμε στη Γαλλία καμία τέτοια δυνατότητα χρηματοδότησης, γιατί ο προσανατολισμός της αποταμίευσης δεν είναι ο κίνδυνος. Και σε μια κοινωνία, στα πλαίσια της οποίας το απρόβλεπτο και το αβέβαιο κυριαρχούν, ποιος έχει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη για να επενδύσει σε πολιετή βάση σε συγκεκριμένες θέσεις. Η αποταμίευση των πολιτών, που σε κάποιες χώρες είναι πολύ ισχυρή, προσανατολίζεται προς συστήματα εγγυημένα, όπως ε, το, ε, το βιβλιάριο ταμιευτηρίου Α στη Γαλλία, που δίνουν λίγα, λίγη απόδοση, αλλά διασφαλίζουν το κεφάλαιο και το κράτος χρησιμοποιεί την αποταμίευση αυτή ε, σε χρήσεις που θεωρεί αυτό ότι είναι χρήσιμες και όχι προς τις μικρομεσαίες. Λοιπόν, η απάντηση δεν είναι εύκολη και αυτό το οποίο λείπει είναι η εμπιστοσύνη. Αν οι αποταμιευτές και αν οι μελλοντικοί επενδυτές δεν έχουν εμπιστοσύνη, δεν θα ρίξουν τα χρήματά τους στις γαλλικές ή στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μπορούμε να διαβάζουμε τα πάντα, να γράφουμε τα πάντα για τους κινδύνους και τις μελέτες επιπτώσεων, αλλά δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Στη Γερμανία υπάρχουν μεγάλες μικρομεσαίες, στη Γαλλία μικρότερες. Στην Γερμανία είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσα σε μια πολυετή διάρκεια με ίδια κεφάλαια. Σήμερα λοιπόν το θέμα το οποίο τίθεται, για το οποίο δεν έχω απάντηση, είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε την αίσθηση της αγάπης για τον κίνδυνο της επιχειρηματικότητας στους επενδυτές, σταθεροποιώντας τις οικονομίες μας και βρίσκοντας τότε τις προσφερόμενες καταλληλότερες λύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τεμπάκερ Και θα ζητήσω συγγνώμη γιατί θα πρέπει να φύγω κατά τη διάρκεια της ομιλίας για να υποδεχθώ τον προσκεκλημένο μας. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Προσπάθησα να διευκρινίσω στην αρχή της ομιλίας μου ότι δεν υπάρχει, θα έλεγα, μία μικρομεσαία είναι διαφορετικές μεταξύ τους οι μικρομεσαίες και δεν μπορεί να υπάρξει λογική το ένα νούμερο κάνει για όλους. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές στις διαφορετικές κατηγορίες μικρομεσαίων έτσι ώστε οι γνώσεις αυτές να μεταφερθούν σε όλες τις χώρες. Δεύτερον, όταν γράφει κανείς ε, νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν πρέπει να επιβαρύνουμε επιπλέον την κατάσταση και ιδιαίτερα το, τις μικρομεσαίες ε, στις ε, απαιτήσει σε επίπεδο κεφαλαίου και όλες οι απαιτήσει που χρησιμοποιούνται, που ε, ισχύουν για τη λειτουργία των τραπεζών, όλα αυτά δείχνουν τον σημαντικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από ό,τι φαίνεται η χρηματοπιστωτική βιομηχανία σήμερα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διανέμεται το κεφάλαιο και αυτό θα επηρεάσει εκ νέου τις μικρομεσαίες αρνητικά. Έγινε μία παρατήρηση επίσης σχετικά με την πολυδιάσπαση των χρηματοπιστωτικών ε, αγορών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε οριακές καταστάσεις ε, δημιουργούνται τεράστιες διαφορές στο ύψη των επιτοκίων η ενημέρωση για υπάρχοντα προγράμματα προς τους επιχειρηματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κάτι το απαραίτητο. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Έχουμε κάνει πολλά προγράμματα τα οποία τρέχουν, αλλά θα πρέπει να ενταθούν και να συνεχιστούν. Τώρα για την εσωτερική αγορά και την έννοια του κινδύνου η οποία εξαφανίζεται από τις αγορές αυτές. Πολλοί ε, διασώζουν πολλά χρήματα γιατί φυσικά ε, δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν τις επενδύσεις τους, αλλά από την άλλη όμως ε, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εξ αυτού προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ε, χωρών να δώσουν κίνητρα είτε φορολογικά είτε άλλου τύπου έτσι ώστε οι χρηματοδοτήσεις να συνεχίσουν να ρέουν και οι αποταμιεύσεις να μην μένουν αδρανείς. Περιμένω τα σχόλιά σας, θα συναντηθώ περαιτέρω μαζί σας και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Ντεμπάκερ να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 18η Οκτωβρίου. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει την 28η και 29η Νοεμβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας αναμένεται για την 17η ή 18η Δεκεμβρίου και η τελική ψήφος τον Φεβρουάριο ε, του 2013. Σε λίγη ώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα την ακρόαση δηλαδή με τον κύριο Ντράγκη ε, ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς σχεδόν στο ωράριό μας, στη σωστή ώρα. Θα ήθελα και πάλι να χαιρετήσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Μάριο Ντράγκη. Δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσω φυσικά σε εσά. Σήμερα το πρωί θα αναφερθεί σε εμά σε αυτή τη δημόσια ακρόαση υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο νομισματικός διάλογος και σας παρακαλώ να κρατήσετε χωριστά τα ερωτήματά σας στις δύο αυτές ενότητες. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστηματικού Κινδύνου. Λοιπόν, χωρίς καμιά άλλη περιστροφή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Σάρων, αγαπητοί και έντιμοι βουλευτές. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπορώ να ευχαριστώ ενώπιον τη Επιτροπή σας σήμερα για να σα πληροφορήσω σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο αυτό συμπληρώνει την τεχνογνωσία που έχουν οι κεντρικέ τράπεζες και οι εθνικοί επόπτες και φυσικά και οι ευρωπαϊκές εποπτικέ αρχέ με το να δίδει αυτό το οποίο έχει γίνει ως γνωστό, γνωστό ως οι μακρο, μακροποπτικές ε, προοπτικές. Ο ρόλος του λοιπόν είναι να αντιμετωπίζει τους κινδύνους σε διάφορους τομείς και να βλέπει τα τροτά σημεία, ιδίως στον τραπεζικό τομέα και να εξετάζει και σε γενικότερο επίπεδο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τους μεσοπρόθεσμους κινδύνους. Επί τη βάση αυτής της ανάλυσης, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με προσπάθειες ε, διορθωτικών δράσεων, το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έχει στόχο να προστατεύσει την ευρωπαϊκή οικονομία από την ευθραυστότητα και την τροτότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Ένα σημαντικό βήμα στο ρόλο του Συμβουλίου αυτού ήταν η δημοσίευση του πρώτου κατά κάποιο τρόπο πίνακα ε, κινδύνου το Σεπτέμβριο του 2012. Ο πίνακας αυτός αξιολόγησης, γνωστός ως dashboard, ήταν μια αίτηση του Κοινοβουλίου μέσα στα πλαίσια της ε, νομοθετικής διαδικασίας που οδήγησε στη δημιουργία του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Αποτελείται από μια σειρά ποσοτικών τε και ποιοτικών δικτών που έχουν σαν στόχο να ποσοτικοποιήσουν και να εντοπίσουν το συστημικό κίνδυνο. Το dashboard αυτό, ο πίνακας ελέγχου έχει δημιουργηθεί με συνεργασία και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Είναι μία από τις βασικές πηγές πληροφορίες που συζητά το Ευρωπαϊκό Συστημικό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει τροτά σημεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης. Ο πίνακας ελέγχου θα την χάνει τριμηνίας επιχειροποίησης και κοιτάζει έξι κατηγορίες κινδύνου και κατατομής και εγκάρσια σε όλο το χρηματοπιστωτικό τοπίο. Θα πρέπει να θεωρηθεί λοιπόν ένα βασικό στοιχείο πληροφόρησης το οποίο μπορεί να κατευθύνει περισσότερο τις περαιτέρω αναλύσεις συστημικού κινδύνου. Αλλά δεν είναι ένα πλήρες σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να δημοσιεύει αυτό τον πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία που περιλαμβάνει στην ε, ιστοσελίδα του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Έρχομαι τώρα στην τωρινή συγκυρία. Η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και το χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζουν ακόμα προκλήσει και είναι κεφαλαιώδε να έχουμε υπόψη μα τα προβλήματα που προέρχονται από το συστημικό κίνδυνο. Υπάρχουν όμω λόγοι μεγαλύτερης εμπιστοσύνη με την προπόθεση ότι οι λήπτε αποφάσεων θα συνεχίσουν να εφαρμόσουν τα συμπεφωνηθέντα μέτρα με αποφασιστικότητα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει μεγαλύτερη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Συμπεριλαμβάνουν επίσης συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις για να είναι ανθεκτικότερες ή ανθεκτικότερα και καλύτερα λειτουργούντα τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και επίσης και η ανάπτυξη ενός θεσμικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από μακροεποπτική προοπτική υπάρχουν τρεις κέρι και κύριοι κίνδυνοι. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι υπαναχωρήσεις στην εφαρμογή συμπεφωνημένων μέτρων. Δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξουν προβλήματα στις τράπεζες σε ό,τι αφορά την κερδοφορία τους και τη λειτουργία τους. Και τέλος υπάρχουν βρόχοι ανάδρασης μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την παροχή πίστοσης που τελικά θα έχει επιρροή και στην πραγματική οικονομία. Το να ανανεώσουμε την παροχή πιστώσεων είναι σημαντικό και κέριο για την ανάκαμψη παρά το γεγονό ότι έχουν μειωθεί οι εντάσει στην αγορά, η χρηματοοικονομική δραστηριότητα έχει πληγεί και παραμένει σε χαμηλό επίπεδο σε πολλά σημεία του συστήματο. Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλο τη μακροπροληπτική πολιτική είναι η ανάκαμψη τη εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Για να μπορέσει κανεί να εξασφαλίσει αυτή την εμπιστοσύνη των επενδυτών στι τράπεζε, είναι απαραίτητο να υπάρχει και κάποια καλύτερη διαβεβαίωση για την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών φορέων. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τις αρχές. Καταρχήν, μία επιλογή είναι να υπάρχει μεγαλύτερη αποκάλυψη σε σχέση με το επίπεδο αποθεμάτων. Δεύτερη ε, επιλογή είναι εποπτικός έλεγχος της ποιότητας των αποθεματικών και με έλεγχο ομοτήμων ενδεχομένω και με εκτίμηση από τρίτου φορεί. Και μια τρίτη επιλογή, όπου είναι απαραίτητη, είναι το να δημιουργηθούν και χωριστοί φορεί οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν στοιχεία ενεργητικού χαμηλή ποιότητα. Το σημαντικό <clears throat> έργο αυτό ήδη γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για να εξασφαλίσει την αντοχή του τραπεζικού τομέα, να προωθήσει τη δημιουργία στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας και για την εναρμόνιση των βασικών παραμέτρων όπως είναι τα δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται. Το Συμβούλιο επίσης θα υποβάλει και περαιτέρω προτάσει για τη μακροπροληπτική πολιτική, ιδίως για τα τροτά σημεία που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Εν όψη λοιπόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένε αγορέ πίστη, το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου μαζί με την Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει προσκόμματα και εμπόδια σε ό,τι αφορά ορισμένα προϊόντα, όπως είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και τις ανταλλαγές πιστοτικής αθέτησης. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε τους κινδύνου που προέρχονται από αυτές τις ενέργειες και θα σας παρουσιάσω την πρόοδο και τα θέματα αυτά στο, στην επόμενη ακρόαση στο πρώτο εξάμεινο του 2013. Η εξέταση από το Συστημικό Συμβούλιο του Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Χώρου ξεπερνάει το τραπεζικό και μονοτομέα. Σήμερα θέλω να εστιάσω περισσότερο στο θέμα των κεντρικών αντισυμβαλωμένων και των ε, ομολόγων που είναι σε διαπραγμάτευση εκτός αγοράς, over the counter δηλαδή στα Ρωμαϊκά. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το ρόλο που έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στην παροχή συμβουλών στα θέματα αυτά. Η εφαρμογή των προτύπων των G20 για την κεντρική εκαθάριση με κεντρικού αντισυμβαλωμένου όλων των ομολόγων εκτό αγορά έχει σημαντικέ επιπτώσει για όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου άρχισε να εξετάζει τι συστημικέ ε, συνέπειες του πιο σημαντικού ρόλου των κεντρικών αντισυμβαλωμένων που θα παίξουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο μέσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η μακροπροληπτική εξέταση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων περιλαμβάνει ιδίω την ε, υπερκυκλική ε, λειτουργία των ε, κουρεμάτων και των περαιτέρω δραστηριοτήτων που μπορούν να λάβουν χώρα στην αγορά πίστης. Αυτά μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην αγορά. Επίσης, η ο κίνδυνος αντισυμβαλωμένου, ο οποίος μειώνεται από τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους, παράλληλα συνοδεύεται από μια αύξηση του κινδύνου που επέχουν οι ίδιοι κεντρικοί αντισυμβαλωμένοι. Επομένως, θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η συστημική αντοχή αυτών των κεντρικών αντισυμβαλλομένων για την εκαθάριση των ομολόγων. Σε ό,τι αφορά τις εγγύησεις, το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έχει, έχει συμβουλεύσει την Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει την αντοχή των κεντρικών αντισυμβαλωμένων με καλύτερο ορισμό των επιλέξιμων εγγύησεων και του πλαισίου στο οποίο ορισμένε εγγύησεις μπορούν να γίνουν δεκτές από τους κεντρικού αντισυμβαλωμένου. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου επίσης έχει δώσει συμβουλές ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι λόγω διασταυρούμενων εγγύησεων και να ληφθούν υπόψη για την εκαθάριση μεταξύ μη χρηματοπιστωτικών φορέων που λειτουργούν στις αγορές παραγωγών, το Συμβούλιο έχει προτείνει να μειωθεί η δυνατότητα για αυτές τις επιχειρήσεις να συμψηφίσουν εκτός των ε, κεντρικών αποθετηρίων ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ο οποίος προέρχεται από τον κίνδυνο συμβαλωμένου. Δυστυχώς αυτό δεν αντιμετωπίζει πλήρως τις, ε, τα τροτά σημεία τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί από το Συστημικό Συμβούλιο και λόγω αυτών των ε, στοιχείων δεν έχει μπορέσει η Συμβουλή του Συστημικού Συμβουλίου να μεταφραστεί, να μεταφραστεί πλήρως σε νέα πρότυπα οι αγορές ομολόγων εκτός ε, οργανωμένων αγορών έχουν να αντιμετωπίσουν κινδύνους που προέρχονται από πρακτικές της αγοράς που έχουν γίνει ιδιαίτερα ε, διαδεδομένες στο λεγόμενο σκιώδη τραπεζικό τομέα. Παραδείγματος χάρη, εγγυήσει που δίδονται από ένα πελάτη μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν από τον δανειστή για τις δικές του ανάγκες δανειοδότησης. Αυτή η εκ νέου ενυποθήκευση μπορεί να αφορά πολλές φορές το ίδιο στοιχείο εγγύησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί μια αλυσίδα μόλυνσης σε εισαγωγικά εάν οποιοδήποτε συμβαλόμενο δεν τηρήσει τα υπεσχημένα. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν τα, οι εγγύησει ε, εκπροσωπούνται από ρευστό χρήμα, το χρήμα αυτό μπορεί να επανεπενδυθεί από τον δανειστή. Και εάν αυτή η επανεπένδυση γίνει σε ε, επισφαλή στοιχεία ενεργητικού με μεγάλη διάρκεια λήξης δημιουργείται ο λεγόμενος κίνδυνος ανασφάλειας σε σχέση με τα, με τα στοιχεία αυτά ενεχείρου. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου έχει επίση αντιμετωπίσει τα νέα σχέδια για την Τραπεζική Ένωση και χαιρετίζει ιδιαίτερα την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Είναι σαφέ ότι τα μακροπροληπτικά ωφέλη ενό ενιαίου μηχανισμού ελέγχου θα ενισχυθούν αν υπήρχε ένα επαρκές κοινό σύστημα επίλυσης για τις τράπεζες χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Οι πρωτοβουλίε τη Κομισιόν για τη δημιουργία ενό ενιαίου μηχανισμού επίλυση για τραπεζικού οργανισμού και για τον συντονισμό τη χρήση των εργαλείων επίλυση μέσα σε μια τραπεζική ένωση είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το ενθαρρύνουμε. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου εξετάζει τι επιπτώσει της ε, την, ε, τις προτάσεις του, για το λεγόμενο SSM, τον, απλό, τον ενιαίο μηχανισμό ε, ασφάλειας. Αυτό επηρεάζει και την μακροπροληπτική πολιτική. Το να έχει, το να υπάρξει μία ε, ενιαία εξουσία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να δημιουργεί από θέματα ασφαλείας αντικυκλικού χαρακτήρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους προ... μακροπροληπτικούς κινδύνους, όπως αναφέρεται και σε νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο συστημικού κινδύνου έχει τονίσει ότι η μακροπροληπτική πολιτική πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη για να μπορέσει να εμποδίσει την ενίσχυση των συστημικών κινδύνων. Οι λήπτε αποφάσεων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, να αντιμετωπίσουν και να καταπραίνουν του κινδύνου από τη στιγμή που εντοπίζονται και όχι να, να παραμείνουν στα πλαίσια τη αδράνεια. Η ευκαμψία μπορεί να αντισταθμιστεί από την δυνατότητα των μέτρων να μειώσουν τις, ε, τα αποτελέσματα εξωτερικοτήτων που δεν γίνονται αντιληπτές. Είναι απαραίτητο λοιπόν να συνεχίσουν οι προσπάθειες για μια πιο έντονη μακροπροληπτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρώτα αποτελέσματα μπορεί να αναμένονται στον επόμενο χρόνο. Συγχρόνω, η οργάνωση του ίδιου του Συστημικού Συμβουλίου και οι προσπάθειες που καταβάλλονται από αυτό θα ενισχυθούν το 2013. Τρία μέλη της Διευθύνουσα Επιτροπή του, του Συστημικού Συμβουλίου, ο Στέφαν Ίγκλης, ο Αντρέ Σαπίρ, ο οποίο είναι επικεφαλή τη Επιστημονική Επιτροπή και ο Βίτορ Κωνσταντσιο, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα, εξετάσουν τη λειτουργία του Συστημικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη και το, την προοπτική της επικείμενης Τραπεζικής Ένωσης. Εργαζό, εργάζεται το Συμβούλιο επίσης για την εφαρμογή του μηχανισμού δράση ή εξήγηση, act or explain, ώστε να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν σωστές ανταποκρίσεις στις συστάσεις του Συστημικού Συμβουλίου. Οι πρώτες συστάσεις του Συστημικού Συμβουλίου που διατυπώθηκαν το 2011 έχουν εκπνεύσει μέσα στο 2012. Επομένως, ο μηχανισμός Actor Explain, πράξε ή εξήγησε, έχει λειτουργήσει σωστά, συγχρόνως. Έχουμε πολύ έργο μπροστά μας για να βελτιώσουμε το πλαίσιό μας για αξιολόγηση. Η Γραμματεία του Συστημικού Συμβουλίου έχει έρθει σε επαφή με εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς με διεθνείς φορείς όπως είναι το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, ο, ΟΣΑ και τα λοιπά για να μπορέσει να αποκομίσει στοιχεία από την εμπειρία τους. Εν κατακλείδη θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι πολύ σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην κατανόηση των συστημικών κινδύνων και στο σχεδιασμό των μακροπροληπτικών πολιτικών μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την ενεργή συμμετοχή και την προσήλωση όλων των επιτροπών και φορέων του, συστημικού, του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. <clears throat> Με την ευκαιρία της αλλαγής της Προεδρίας της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μάρτιν Χέλβικ, τον πρώτο πρόεδρο αυτής της Επιτροπής και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στο μέλλον, όπως και στον Αντρέ Σαπίρ που αναλαμβάνει αυτή την Προεδρία. Κατανοώ, θα έχετε την ευκαιρία να ανταλλάξετε απόψη με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο αυτής της Επιτροπής εν καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαι τώρα στη διάθεσή σας για ερωτήματα. Um, ευχαριστώ πολύ. Ως συνήθως Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε δέκα ερωτήσεις προς τον κύριο Ντράγη. Έχουμε κατανείμει τον χρόνο και τους ομιλητές σύμφωνα με τον κανόνα αντεχών φυσικά. Για να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερο τον χρόνο θα πάρω τις ερωτήσεις κατά ομάδες γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Πρώτοι τρει θα είναι Χούμπνερ, Φερέρ και Σμιτ. Η κυρία Χούμπνερ που είναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι για την πρόληψη αλλά και την διασπορά του κινδύνου απαιτούνται μηχανισμοί εποπτείας. Πράγματι οι συστημικές αυτές, ε, ε, τα συστημικά σημεία ευθραστότητας ε, των τραπεζών ιδιαίτερα δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και σταθερό, είναι κάτι το οποίο αλλάζει και θα πρέπει να προσαρμόσουμε και τον τρόπο που προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Ελπίζουμε ότι ελπίζουμε μάλλον ότι ο μηχανισμός αυτός θα μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς επιμέρους μικρότερους μηχανισμούς και δεν θα οδηγήσει στην διαίρεση της εσωτερικής αγοράς σε ε, τράπεζες και πιστοτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ και αντίστοιχα εκτός ζώνης ευρώ. Τα κριτήρια τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εντοπισμό των συστημικών κινδύνων σε σχέση με την έκθεση των επιχειρήσεων είναι ανεπαρκή. Δεύτερον, θα ήθελα να μάθω αν πιστεύετε ότι η διέρεση του, ε, της εσωτερικής αγοράς ανάμεσα σε ζώνη ευρώ και εκτός Ζώνη ευρώ θα αποτελέσει ένα επιπλέον συστημικό κίνδυνο. Και χωρίς μηχανισμό επίλυσης των προβλημάτων πώς βρίσκετε εσείς ότι θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστά τον κίνδυνο. Η κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. τα δάνεια τα οποία δίδουν τα πιστοτικά ιδρύματα είναι ε, κάτι το οποίο πλέον έχει καταστεί τρομακτικό πρόβλημα στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Δεν υπάρχει ροή δανειοδότησης, πάρα πολύ απλά. Το θέμα έχει τεθεί εδώ ε, και ακόμα και οι βιώσιμες επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να παίρνουν δάνεια. Και ακόμα μάλιστα και χειρότερο αυτό από τράπεζες οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από το δημόσιο δεν δίδουν, δεν μεταφέρουν τα χρήματα στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι ε, τρομακτικό συστημικό κίνδυνο. Δεύτερο θέμα. Ο, μακρο, ε, μακροελεγκτικός, ε, η μακροελεγκτική εποπτεία, η προληπτική εποπτεία. Το Συμβούλιο έχει, Κινδυνού έχει κάνει κάποιες συστάσεις για τα θέματα της λιτότητας Αναρωτιέμαι όμως αν οι συστάσεις αυτές εφόσον εφαρμοστούν τι συνέπειες θα έχουν για χώρες όπως η δική μου, η Πορτογαλία, οι οποίες εφαρμόζουν τις προτάσεις και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και ε, ε, οδηγεί επίσης σε μια τρομερή ύφεση και σε επιπλέον μέτρα λιτότητας. Και τελικά αυτό είναι ο κίνδυνος για χώρες σαν τη δική μου. Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Η ερώτησή μου συνδέεται με την ερώτηση που έθεσε η κυρία Χίμπνερ. Τι θα συμβεί στην περίπτωση κατά την οποία πολλές χώρες και τράπεζες βρεθούν εκτός ε, πιστοτικής ένωσης, εκτός τραπεζικής ένωσης και τι θα γίνει με την επίβλεψή τους και με την εποπτεία τους. Ε, σας έχω ενοχλήσει τον τελευταίο καιρό σε σχέση με το λεγόμενο χάσμα των φύλων. Έχετε το ίδιο πρόβλημα και στην ε, Κεντρική Τράπεζα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια δυνατότητα σταθεροποίησης επιπλέον όταν μόνο άνδρες ασχολούνται με την νομισματική πολιτική στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει και μια επιστολή από έναν πολύ γνωστό οικονομολόγο που λέγει ότι το να αποφασίζουν μόνο άνδρες για τέτοια θέματα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και αυτό το οποίο κάνετε κύριε Πρόεδρε είναι μέχρι τώρα εξαιρετικό, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα με την εκπροσώπηση των δύο φίλων σε αυτό το επίπεδο. Καλώς λέει Πρόεδρος, ο κύριος Ντράγκη. Έχετε 7 λεπτά για να δώσετε απαντήσεις στις ερωτήσεις. Um, me, uh, now on the criteria for identifying τα κριτήρια για τον, για τον εντοπισμό των συστημικών προβλημάτων. Εμείς έχουμε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια καλή βάση συζήτησης. Καταρχάς, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Χρησιμοποιούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαν μια πλατφόρμα για να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Νομίζω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε στο ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι το FSB εδώ και 3-4 χρόνια είχε ήδη εντοπίσει κάποια κριτήρια τα οποία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν για την καταλογοποίηση ε, των συστημικά σημαντικών οργάνων. Ε, φυσικά, ε, εμεί λειτουργούμε σαν σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα για τη ζώνη ευρώ. Οπότε Υπάρχουν λοιπόν κάποια ιδρύματα πιστοτικά τα οποία είναι συστημικά ή θεωρούνται συστημικά σε επίπεδο ευρώ αλλά όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε στους καταλόγους τους οποίους συντάσσουμε. Λοιπόν, τέθηκαν επίσης δύο ερωτήσεις για το εάν ο ενιαίος προληπτικός αυτός εποπτικός μηχανισμός θα σπάσει την αγορά ανάμεσα σε μία αγορά ευρώ και σε μία αγορά εκτός ευρώ. Δύο πράγματα να πω εγώ. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε και εξετάζουμε το SSM μέχρι τώρα είναι ανοιχτός και για τις χώρες εκτός ευρώ που θέλουν να συμμετέχουν. Εμείς θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να συμμετέχουν είναι τέτοιες που να ταυτίζονται με τις συνθήκες μέσα στις οποίες κινούνται οι χώρες ευρώ. Και θέλουμε αυτό να είναι συμβατό και με την νομική βάση η οποία στηρίζει και βρίσκεται κάτω από το SSM. Η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σαφεστάτη. Είμαστε εμείς υπέρ της ισοτιμίας μελών εντός και εκτός ζώνης ευρώ. Για την εσωτερική αγορά δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο ρόλος του EBA θα διευκολυνθεί. Θα διευκολυνθεί από ένα ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, εν λειτουργία μηχανισμό, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι ο, ο, ο κανόνας αυτός, ο ενιαίος, θα εφαρμοστεί από ένα μεγάλο, μεγάλο ποσοστό των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι η εσωτερική αγορά θα ωφεληθεί από τον ενιαίο ελεγκτικό μηχανισμό. Φυσικά θα πρέπει να βρούμε τις πρακτικές και τις διαδικασίες και τις μεθόδους που θα το πετύχουμε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η εσωτερική αγορά θα βελτιωθεί από τις εξελίξεις αυτές και δεν θα βλαφθεί από αυτές. για την δυνατότητα που μπορεί να υπάρξει ε, να λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός ο ελεγκτικός ο ενιαίος χωρίς να φυγούν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία γιατί τμήμα ακριβώς αυτών των μηχανισμών των ελεγκτικών μακροπρόθεσμα ε, είναι η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες εποπτικές αρχές. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει και στον τομέα της Τραπεζικής Ένωσης. Να μην ξεχνάμε πως έχουν ιστορικά, θα έλεγα, ξεκινήσει αυτές οι εποπτικές αρχές και αρχές επίλυσης διαφορών. Uh, Λογική είναι να μην χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων στην περίπτωση κατά την οποία δημιουργηθεί πρόβλημα με μία τράπεζα. Να μην χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων και δεν θα πρέπει να υπάρξει και διάλυση του συστήματος ε, πληρωμών. Δυστυχώς κάτι τέτοιο συνέβη και στις δύο περιπτώσεις ε, με, τις, με τους Lehman Brothers. Είχαν συμβεί προβλήματα αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές χώρες και πριν από την περίπτωση της Lehman Brothers. Πάντως, το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι να αποφύγουμε περαιτέρω κινδύνους. Αν μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος δεν θα επιτρέπει ε, να οδηγούνται στην αποτυχία ε, μεγάλα πιστοτικά ιδρύματα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε τα προβλήματα. Να μην χρησιμοποιούμε λοιπόν τα χρήματα των φορολογουμένων και να διασφαλίσουμε έτσι ώστε το σύστημα πληρωμών, το σημαντικότερο κομμάτι του χρηματοδοτικού συστήματος να συνεχίσει να λειτουργεί. Προβλήματα θα δημιουργηθούν. Αρκετές τράπεζες μπορεί να κλείσουν, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να διακοπεί το σύστημα πληρωμών. Έχουμε διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικούς κανόνες σε διαφορετικές χώρες γύρω από όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς αυτή η αρχή ε, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να περιορίσει τη διασπορά των αρνητικών συνεπειών προβλήματος σε ένα πιστοτικό ίδρυμα και έτσι θα τονίσει την εμπιστοσύνη προς το ευρωπαϊκό σύστημα. Τώρα για την, για την ύφεση και τους κινδύνους που παρουσιάζει η ύφεση. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαδικασία της εξυγίανσης, της δημοσιονομικής βάχη πρόθεσμα θα πιέσει και θα συρρυκνώσει την παραγωγή σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τι είναι όμως εναλλακτικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να μην ξεχνάμε ότι η κρίση ξεκίνησε από μια αποστροφή στον κίνδυνο που αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα όπως ε, η τα μη βιώσιμα ποσοστά χρέους σε πολλές χώρες της Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε και πρέπει να το διορθώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να είμαστε σύντομοι και αποτελεσματικοί. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό βασιζόμενοι στις αρχές φυσικά της κοινωνικής δικαιοσύνης, αυτό είναι μια σαφεστάτη απέτηση και θα πρέπει να το πετύχουμε όπως έχω επανειλημμένα πει ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει πλέον μια προοπτική μια προοπτική σε εθνικό επίπεδο αποκατάστασης της ανάκαμψης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αυτή είναι η ελπίδα. Η διαδικασία αυτή είναι αναπόδραστη. Τέλος, για το θέμα των διαφορών στα δύο φύλλα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο κύριε Σμιτ. Είναι σαφές. Τα στοιχεία είναι υπερημών αν δείτε τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα με τη χρηματοπιστωτική κρίση, μόνο άνδρες ασχολήθηκαν με αυτήν. Έχετε λοιπόν απόλυτα δίκιο, πρέπει ε, γρήγορα να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Δεν θέλω να κάνω αναφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας. Πρέπει να πούμε ότι στη δική μας περίπτωση, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή κρίσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί το κενό που έχουμε στο Συμβούλιο. Αλλά θα πρέπει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσπαθήσουν και να βρουν μια κάποια λύση στο θέμα της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών. Πρέπει να σκεφτούμε και να δράσουμε. Το να εκφράζει κανείς σκέψεις χωρίς δράση δεν οδηγεί ε, πουθενά. Πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να το πράξουμε. Ε, σχόλια χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγονται από τη διαμηνία Κύριε Δράκη ναι, αυτά που λέτε, αλλά τα, αυτό που δεν άκουσα καθόλου από εσά είναι λύσεις. Εντοπίσατε τα προβλήματα, αλλά δεν προτείνετε λύσεις. Για το δανεισμό τίτλων ε, και τις υποθήκες του συστημικού κινδύνους που αυτά προκαλούν. Λοιπόν, δύο σύντομα ερωτήματα για το ποσοστό leverage. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί λένε ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ε, λόγο ιδίων προς ξένα κεφάλαια, μια τέτοια μόχλευση, ε, πολύ περισσότερο. Την προηγούμενη εβδομάδα το είπατε. Ποια θα είναι η αρχιτεκτονική. Δηλαδή εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι διατηρώντας ε, τις εμπορικές και τις λαϊκές τράπεζες με τους ίδιους ε, κανόνες ε, μπορούμε να αποφύγουμε συστημικό κίνδυνο και να αποφύγουμε να περάσει ο κίνδυνος από τη μία περίπτωση στην άλλη. Μήπως κινδυνεύουμε να καταλήξουμε στο αντίθετο. Περιμένω να μου πείτε τη σκέψη σας. Ο επόμενος είναι ο Ήβο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνοντα υπόψη μας κύριε Πρόεδρε, τα όσα κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Σύστημα, δεν νομίζετε ότι θα είχε περισσότερο νόημα να χρησιμοποιήσουμε το Συμβούλιο αυτό και όχι την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να δημιουργηθεί από εκεί ο ενιαίος αυτός μηχανισμός εποπτείας γιατί μεταξύ άλλων θα μπορούσαμε έτσι να είχαμε διάκριση ανάμεσα στην εποπτεία και την νομισματική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα είχαμε και καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι οποίες αποτελούν ε, μέρος του γενικότερου εποπτικού συστήματος προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα εποπτείας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο Νίκος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά, στα μέτρα αντιμετώπισης συστημικού κινδύνου εντάσσεται και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής σε ορισμένες χώρες, καθώς το πρόβλημα ξεκινούσε από τη μη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους ορισμένων χωρών. Αυτό βέβαια φέρνει την ύφεση, το παραδεχτήκατε. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω και που έχει και μια επικαιρότητα είναι το ελληνικό χρέος παρά τα μέτρα αντιμετώπισης συστημικού κινδύνου όπως τουλάχιστον κατάλαβα εννοείται τα, προγράμματα προσαρμογής. Δεν είναι βιώσιμο. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν διάφοροι αναλυτές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σήμερα κάνει δυσμενείς προβλέψεις. Και η ερώτηση δική μου είναι, το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ξεχνώ και την ιδιότητά σας, τι εκτίμηση κάνετε για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους που προβλέπεται σύμφωνα με τις αισιόδοξες προβλέψεις να πάμε στο 120% δεν φαίνεται το 2020. Και αν προβλέπετε ότι δεν είναι βιώσιμο, τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε αφού διαπιστώνετε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα. Δηλαδή θα προτείνετε ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών απευθείας από το μηχανισμό, σκέφτεστε να μην ζητήσετε ολόκληρη την ονομαστική αξία των ομολόγων που έχει αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιτέλους τι σκέπτεστε για να αντιμετωπίσετε έτσι όπως φαίνεται ένα συστημικό κίνδυνο που τα ήδη μέτρα που έχουν ληφθεί δεν τον αντιμετωπίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ευχαριστώ. Όσον αφορά την επανυποθήκευση, επιτρέψτε μου να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτό είναι ένα παλιό πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα το ότι αποτελεί δηλαδή ένα από τα κανάλια προβλήματος μετά από τη Λίμαν. Είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώς και σε ένα βαθμό τουλάχιστον δεν το προσέξαμε ως όλα προβλήματα. Όμως είναι παρόν το ασχολούνται. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με, με τις ναι, εγγύσεις ναι. και την ε, ενεχείρεση. Α, να ξέρετε ότι διάφορες ε, πλευρές φροντίζουν αυτός ο οποίος το κάνει, μετά θα μπορέσει να βρει πίσω αυτά που έχει βάλει. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου επικεντρώνεται στα εξή. Κατά πόσο αυτή η επανεγχειρίαση χρησιμοποιείται σε βάρος ή χρησιμοποιείται για δανεισμό, για ανάγκες δανεισμού. Έπειτα να δούμε πώς το ρευστό χρησιμοποιείται από τον δανειστή και ποια είναι η σχέση των τραπεζών και των μη τραπεζών από μια τέτοια πρακτική. Πώ επίση θα βελτιώσουμε την ενημέρωση και τον έλεγχο τέτοιου είδου συναλλαγών. Δηλαδή, αυτό που μα ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η διαφάνεια. Διότι πρόκειται για ένα από τα μαύρα κουτιά που έχουμε στι δημοσιονομικέ συναλλαγέ. Δηλαδή, το πιο βασικό είναι να μάθουμε περισσότερα για τέτοιε πρακτικέ. Να είναι πιο ορατέ λοιπόν αυτέ οι δράσει. Κάτι το οποίο θα μα διευκολύνει επίση να εντοπίζουμε πιο έγκαιρα του κινδύνου που προκαλούνται από τέτοιε πρακτικέ. Θέλουμε επίσης αρκετές πληροφορίες για να αξιολογούμε τους κινδύνους αυτούς. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για να σχεδιάσουμε και τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Δύο πράγματα σκεφτόμαστε. Πρώτο να βελτιώσουμε τον έλεγχο και την ενημέρωση και το δεύτερο είναι να δούμε τι μέτρα πολιτικής χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε βέβαια καταλήξει το να απαγορεύσετε την πολυεπίπεδη επανεγχειρίαση, αυτό το σκέφτεστε. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Δεν το αποκλείω, αλλά πάντως δεν λέω ότι θα το κάνουμε. Δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά στην σκέψη μας για να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο αξιολόγηση ακόμα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε να μπορέσω να σας πω περισσότερα πάνω σε αυτό. Έρχομαι τώρα στο ποσοστό μόχλευσης. Γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα κάποιο επίπεδο μόχλευσης. Είναι σημαντικό. Μια, ένα από τα δάγματα που πήραμε από την κρίση είναι ότι πολλές ε, τράπεζες θεωρούσαν ε, ρευστό κάτι το οποίο δεν ήταν ρευστό. Και χωρίς να είμαστε κινησιακοί νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό και πρέπει να σταθμίσουμε κάπως αυτό το ποσοστό μόχλευσης σε τέτοια επίπεδα που να μην είναι αντιπαραγωγικό, να μην εμποδίζει τις διατραπεζικές συναλλαγές. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν λειτουργούν καλά αυτές είναι ακριβώς ότι οι ρυθμίσεις για την ρευστότητα έχουν σαν αποτέλεσμα να κοστίζει πάρα πολύ το να δανείζουν χρήματα οι τράπεζες και να δανείζεται κανείς χρήματα από τις τράπεζες. Γι' αυτό και πρέπει να αξιολογήσουμε τις κυκλικές συνθήκες. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να φτιάξουμε buffers και πρέπει να δούμε επίσης τις συνέπειες ιδιαίτερα στις διατραπεζικές αγορές. Πρέπει επίσης να αναθεωρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του ποσοστού κάλυψης ρευστότητας. Μίλησε και με τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής Βασιλείας ως ε, πρόεδρος για να δούμε τι αναθεώρηση μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει η σχέση ανάμεσα στην ε, αναλογία κάλυψης ε, ρευστότητος και αυτό που συζητάμε τώρα. Πιστεύω ότι αυτή η διάδραση έχει τις δικές της ε, συνέπειες στην τραπεζική αγορά. Έρχομαι τώρα στην έκθεση Λικάνεν. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι δημοσιεύθηκε πολύ πρόσφατα και λαμβάνουμε γνώση. Αναγνωρίζει ότι δεν υπήρχε επαρκής ε, κεφαλαιακή κάλυψη και ότι ο συστημικός κίνδυνος προκλήθηκε από την στενή διασύνδεση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πάντως, η πρόορη αναγνώριση και η σωστή αξιολόγηση συστημικού κινδύνου αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, διαπιστώσαμε ότι μα λείπα κάποιε πληροφορίε για την αξιολόγηση αυτή και για την διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και όπω επίση και για την ε, ανάλυση των ε, δραστηριοτήτων του. Συνεπώ, συστήνουμε να υπάρξει μια νομική διάκριση ανάμεσα στι ιδιαίτερα επικίνδυνε τραπεζικέ δραστηριότητε από τι καθαρά αποταμιευτικές. Πρέπει να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος στις αποταμιεύσεις, ακόμα και όταν υπάρχει αυτή η διάκριση. Επίσης, αναφέρει τρεις αδυναμίες η έκθεση. Πρώτον, οι ελάχιστε κεφαλαϊκές απαιτήσει της Βασιλείας, που βασίζεται στους κινδύνους δανεισμού της τράπεζας. Δεύτερον, οι κίνδυνοι ρευστότητος, που δεν καλύπτονται από τους κανόνες της Βασιλείας, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί αυτό οδηγεί στο πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να τα εξετάζουμε αυτά, αλλά επιτρέψτε μου να πω και μια γενική παρατήρηση γι' αυτό. Είτε εσείς για το δίκας μιλήσατε και για τον κανόνα Φόλκερ. Η κατάσταση αυτή του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος διαφέρει πάρα πολύ από ό,τι σχή σε άλλα σημεία του κόσμου. Οι δικές μας οι τράπεζες βασίζονται πιο πολύ στις παραδοσιακές δραστηριότητες δανεισμού από ότι οι αντίστοιχες σε άλλα σημεία του κόσμου. Για μένα λοιπόν αυτό ε, απαιτεί μια πραγματική αξιολόγηση της σχέσης ανάμεσα στον δανεισμό αυτών, τον λιανικό και μη λιανικό. Πριν καταλήξουμε σε κάποια μορφή ρύθμισης που σίγουρα θα διαφέρει, στοιχηματίζω σε αυτό, από αυτό που έχουμε σε άλλα σημεία του κόσμου, γιατί οι τράπεζες είναι διαφορετικές αλλού από αυτές που έχουμε εμείς εδώ. Τώρα η ερώτηση γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να υπάρχει διάκριση αυτή ανάμεσα στην νομισματική ε, πολιτική και της, την εποπτεία. Μετά από τη διάσκεψη του Ιουνίου και την απόφαση εκεί να ξεκινήσει αυτός ο μηχανισμός ενιαίας ε, μακροπληκτικής ε, εποπτείας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον ε, συνδέεται με την αρχή αυτή. Σίγουρα η σταθερότητα τιμών είναι το καθήκον μας και μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτό σαν κεντρικό μας μέλημα. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι τώρα δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια στους νομοθέτες για να δράσουν διαφορετικά. Το θέμα είναι στην πράξη πώς θα διασφαλίσουμε ότι η διάκριση αυτή είναι πραγματική. Και εδώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας προσφέρει κάποια εργαλεία, κάποια μέσα για να φροντίσουμε γι' αυτό η δυνατότητα το Συμβούλιο να μπορεί να εξουσιοδοτεί πλήρως για την ε, μακροπροληπτική αυτή εποπτεία, αυτός είναι ένας κανόνας που εξετάζουμε. Και εδώ μπορούμε βέβαια να το ξανασυζητήσουμε, αλλά ο τρόπος που δουλεύουμε με τους εθνικούς επόπτες είναι Τέτοιο που η νομισματική πολιτική μένει εντελώ απ' έξω από τον χώρο εκείνο στον οποίο δουλεύουμε. Οπότε οι εθνικοί επόπτες θα νιώσουν, θα ενστερνιστούν τη διαδικασία αυτή. Δεν πρόκειται να χάσουν από εποπτεία, δεν θα τη δώσουν, θα την παραχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι δικέ τους αρμοδιότητες από την άλλη μεριά δεν αυξάνονται. Αποτελούν μέρος της διαδικασίας λήψη αποφάσεων σε επίπεδο εποπτείας για την Ευρωζώνη. Δεν θα πρόκειται για κάποια εξουσιοδότηση που δίνουμε, θα είναι από κοινού η δράση μας σε αυτή τη διαδικασία. Συνεργαζόμαστε μαζί τους. Και σας το λέω αυτό επίσης ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ επικοδομητικό, να ξέρετε. Ε, δεν υπάρχει καθόλου αμυντική στάση από καμία πλευρά. Για την ελληνική κατάσταση, επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι το μόνο που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της Τρόικα για να αξιολογήσουμε πώς έχει η κατάσταση. Χτες συζητήθηκε στο Eurogroup, θα ξανασυζητηθεί και σήμερα, νομίζω ότι τώρα στο ECOFIN αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της Τρόικα. Στο μεταξύ, είναι σαφές ότι η πρόοδος σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων έχει γίνει αντιληπτή, είναι ουσιαστική. Και είναι επίσης σαφές ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Βλέπουμε πρόοδο, βλέπουμε ότι χρειάζεται παραπάνω δουλειά, αλλά για μια οριστική αξιολόγηση για τα θέματα στα οποία εσείς αναφερθήκατε πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της Τρόικα. Um, Ωραία. Τελευταίος γύρος με τέσσερις ε, <clears throat> ομιλητές. Η κυρία Κράτσα, ο Αντολίν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να αναφερθώ στην, ε, στις ανισότητες ε, δανεισμού των επιχειρήσεων και τους κινδύνους που εγκυμονούν για τον κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς στις χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίες ε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα πρόσφατα, το επιτόκιο που χρεώνουν οι τράπεζες για ένα εταιρικό δάνειο έως 1 εκατομμύριο ευρώ με αποπληρωμή 1 με 5 χρόνια, ένα δάνειο που δίνεται συνήθως σε μικρές επιχειρήσεις, ανέρχεται στο 6,5% στην Ισπανία. Το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 6,24% ε, στην Ιταλία, ενώ στη Γερμανία είναι μόλις 4,04% και στη Γαλλία 4,1%. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Αντολίν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ με απόλυτα την άποψη αυτή ότι το να επαναφέρουμε μία, ναι, μία ισορροπία στην αγορά πίστοσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συστημικός κίνδυνος προέρχεται από την διασύνδεση των πιστοτικών οντοτήτων, αλλά μπορεί να προκληθεί και ένας κίνδυνος όταν υπάρχει και μείωση της διασύνδεσης των πιστοτικών ιδρυμάτων. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια αυξανόμενη ένας αυξανόμενος κατακαιρματισμός της εσωτερικής αγοράς στα χρηματοπιστωτικά, υπάρχει μια μετακίνηση των τραπεζικών καταθέσεων και έλλειψη εσωτερικής αγοράς. Δεν κινείται το κεφάλαιο προς τα εκεί που υπάρχει ανάγκη για κεφάλαιο. Επομένως με τον τρόπο αυτό συσσωρεύονται κίνδυνοι στο ευρωσύστημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει όλο και περισσότερο τους κινδύνους του συστήματος το οποίο βρίσκεται σε στασιμότητα και είναι μπλοκαρισμένο. Υπάρχουν επίσης θυγατρικές εταιρείε που έχουν τις μητρικές του εταιρείε σε κεντρικές ε, ε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους και τη ρευστότητά τους λόγω των εποπτών των κεντρικών αυτών χωρών. Εκεί λοιπόν όταν υπάρχει έλλειψη διασύνδεση, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διαχειριστεί αυτούς τους κινδύνους γιατί προς τα εκεί μετακινείται ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση. Με τις εισόρες λοιπόν αυτή υπάρχουν όλο και περισσότεροι κίνδυνοι οι οποίοι εντοπίζονται και συσσωρεύονται στο ευρωσύστημα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα ευρωπαϊκού χαρακτήρα για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και να μπορέσει να επανα, ε, εδρεωθεί η εσωτερική αγορά και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα σύστημα εποπτείας αλλά και ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ώστε να μην μετακινούνται οι καταθέσεις από μια χώρα που είναι επίσφαλη συνθήκες σε μια χώρα που να είναι μεγαλύτερη ασφάλεια και επίσης χρειάζεται ένα κοινό σύστημα επιλύσεως για να αντιμετωπιστούν αυτό όλα αυτά. Συμφωνείτε κύριε δράκη. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι. είπατε για την ομάδα των τριών, μεταξύ των οποίων και ο Αντρέ Σαπίρ θα αντιμετωπίσουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας στα πλαίσια της επικείμενης Τραπεζικής Ένωση. Πώς βλέπετε τώρα την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και του ενιαίου επόπτη. Ο επόπτης θα βασίζεται στο σύστημα ε, στο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ή θα κάνει τι δικέ του αξιολογήσει. Δεύτερον, είπατε ότι το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου προσπαθεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο σε όλου του τομεί τη αγορά και σε όλα τα στρώματα τη αγορά. Σα περιορίζει βέβαια η συνθήκη στι τράπεζε. Ξέρουμε ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ τραπεζών, αλλά όχι μόνο μεταξύ τραπεζών, αλλά και μεταξύ τραπεζών και άλλων πιστοτικών ιδρυμάτων και μεταξύ του σχιώδου ε, τραπεζικού τομέα και μεταξύ των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών, παραδείγματο χάρη. Έχει νόημα να περιορίσετε τι ενέργειέ σα και τι ενέργειε του ενιαίου επόπτη μονάχα στον τραπεζικό τομέα. Και το τρίτο μου ερώτημα είναι το εξή. Είπατε ότι δεν έχετε πολύ περιθώριο ελιγμών σε ό,τι αφορά τη γενική πολιτική σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου συστημικού κινδύνου. Αλλά με τη νέα Τραπεζική Ένωση θα έχετε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών. Θα προσπαθήσετε λοιπόν να εφαρμόσετε μια γενικότερη πολιτική στα πλαίσια αυτά. Ο Γκέι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τράγκη, ήμουνα πραγματικά εντυπωσιαστή από αυτά που είπατε σήμερα το πρωί σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αντιμετωπίσετε την, το μη βιώσιμο επίπεδο χρέους και τις υψηλές ε, το υψηλό βάρος του δανεισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι πολύ θετικό που το είπατε, θέλουμε να το ακούμε πιο συχνά από σας. Δεύτερον, όταν αναφερθήκατε σε ποιοτικά και ποσοτικά μέτρα σε σχέση με τον πίνακα ελέγχου, τον dashboard. Δεν μπορείτε όμως να έχετε άλλα μέτρα και σταθμά σε μία χώρα και σε μια άλλη χώρα, στη δική μου χώρα, στην Ιρλανδία. Έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα αυτού του ηθικού κινδύνου που αναφέρατε προηγουμένως. Από 20% φτάσαμε περίπου σε 130% σε επίπεδο κρατικού χρέους. Αλλά εξακολουθούμε να έχουμε στον εθνικό ισολογισμό στοιχεία τα οποία δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στον ισολογισμό αν θέλουμε να καταμετρούμε με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα <clears throat> και το χρέος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή εμείς τροχοπεδούμε τα πολύ δύσκολα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για να ελέγξουμε τις ταμιακές ροές με το να μην ε, έχουμε αναδιάταξη των γραμματείων Αγγλο-Ιρλανδικού χαρακτήρα. Θα είναι και τα επόμενα μέτρα πάρα πολύ οδυνηρά, αλλά θα πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να λάβουν χώρα. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να πούμε και σε άλλες χώρες κοιτάξτε υπάρχει μεγάλη οδύνη στην Ιρλανδία και θα πρέπει να κάνουμε κάποιο, κάποια κίνηση για αυτά τα γραμμάτια μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου και για το, τα τμήματα του χρέους τα οποία δεν πρέπει να βρίσκονται στους εθνικούς λογαριασμούς. Θεωρητικά έχετε περίπου τέσσερα λεπτά, οπότε μπορείτε να μπείτε και στο επόμενο τμήμα της συζήτησής μας, λέει η κυρία Μπάουλς. Θα έχουμε πέντε λεφτά διακοπή μεταξύ των <laughs> δύο ακροάσεων. Εγώ δεν κάνω διακοπέ, λέει, στι συνεδριάσει μου η κυρία Μπάουλ. Καλά, λέει ο κύριο Δράγκη. Είχα δύο ερωτήματα σε σχέση με τον κατακαιρματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε ότι έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό. Να πω μονάχα εν συντομία ότι υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τον κατακαιρματισμό αυτό. Ο ένας είναι προσωρινός, το ελπίζουμε τουλάχιστον, ο άλλος είναι διαρθωτικός. Ο προσωρινός είναι κάτι που οφείλεται στην κρίση εμπιστοσύνη η οποία σοβεί στην περιοχή του ευρώ στους τελευταίους μήνες. Εξακολουθεί να ισχύει. Ο δεύτερος λόγος είναι διαρθωτικός και αυτό είναι η σύνδεση μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και των κρατικών οικονομικών. Όταν επιδεινώνονται οι προπολογισμοί σε εθνικό επίπεδο, τότε οι τράπεζε που βρίσκονται στο έδαφο μια χώρα είναι υποχρεωμένε να πληρώνουν περισσότερο για τη χρηματοδότησή του. Αυτό επιβαρύνει την, ε, τα επιτόκια δανεισμού του. Πώ θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Καταρχήν χρειαζόμαστε να υπάρξει από, την εθνική, από τις εθνικές κυβέρνησεις συνέχιση τη προσπάθειας μεταρρυθμίσεων και εδραίωση των δημοσιονομικών του για να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητα με διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις, αλλά χρειαζόμαστε και ένα ε, εργαλείο για να αποφύγουμε τις, ε, τους λεγόμενους κινδύνους ουράς, tail risks, που είναι ο κίνδυνος να αλλάξει, να βγει κανείς και από το ευρώ. Αυτή είναι, αυτές είναι οι λεγόμενες ενέργειες που γίνονται με τις οριστικές πράξεις νομισματικού χαρακτήρα. Ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν το οποίο έχει επινοηθεί και έχει εγκριθεί στη διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, το, την Ευρωπαϊκή Αρχή Επίλυσης και την εγγύηση για τις τραπεζικές καταθέσεις. Εμείς έχουμε ξεκινήσει με το πρώτο θέμα, <clears throat> τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας που θα μας δώσει όταν θα είναι λειτουργικός πλήρως ο μηχανισμός αυτός θα δώσει σε όλους αυτούς που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ και σε αυτούς που είναι έξω από τη ζώνη του ευρώ ε, εμπιστοσύνη στο ότι υπάρχει κεντρική εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών, φυσικά και με τη συμμετοχή των εθνικών εποπτών, αλλά όλων από κοινού. Αυτό από μόνο του θα αυξήσει και την εμπιστοσύνη η οποία αφορά στους ισολογισμούς των τραπεζών. Το δεύτερο στοιχείο είναι το να μπορέσουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή αρχή επίλυσης και μόνο στο τέλος, το τρίτο στοιχείο, είναι η εγγύηση των καταθέσεων. Γιατί, ειλικρινά, αν σας λένε, μπορείτε να αναλάβετε τον κίνδυνο για κάτι το οποίο σας είναι άγνωστο, θα απαντούσατε να το ελέγξω, να δω τι ακριβώς γίνεται, προτού αναλάβω αυτήν την ε, ευθύνη. Και δεν μπορεί κανείς να, κατα, ε, να καταργήσει τους εθνικούς μηχανισμούς εγγύησης καταθέσεων χωρίς να ξέρει περί πρόκειται. Αυτοί οι τρεις πυλώνες θα επαναφέρουν την εμπιστοσύνη, θα σπάσουν το φαυλοκύκλο μεταξύ τραπεζών και κρατικών προϋπολογισμών, αλλά έχουν διαφορετικό χρόνο, χρονικό ορίζοντα ενεργοποίησης. Για να βγούμε λοιπόν από αυτήν την κατάσταση κατακαιρματισμού και συμφωνώ με τη διάγνωσή σας, αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι να αποφύγουμε τα διαφορετικά επιτόκια. Πολλές φορές μια εταιρεία με δύο θηγατρικές, μία σε μια χώρα και μία σε άλλη χώρα μέλους, πληρώνει τελείως διαφορετικά επιτόκια. Υπάρχουν ιστορίες που μια διαμεθοριακή επιχείρηση, η ίδια επιχείρηση, πληρώνει τελείως διαφορετικά επιτόκια σε δύο χώρες. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες ζητούν ένα στεγαστικό δάνειο και είναι τελείως διαφορετικά τα επιτόκια από τη μια μεριά ή από την άλλη μεριά των συνόρων. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος κατακαιρματισμός, έλλειψη ε, και όλα αυτά πάρα πολλοί δείκτες τα καταγράφουν αυτά. Εμείς θα πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση και επίσης τούτου λεχθέντος. Κάποια πράγματα έχουν βελτιωθεί στους τελευταίους δύο-τρεις μήνες. Πιστεύω όμως ότι έχουμε πολύ δρόμο να διατρέξουμε και είναι και ανηφορικός ο δρόμος αυτός γιατί θα πρέπει όλα αυτά τα μέτρα να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν αναφερθήκατε στο ερώτημα. Συγγνώμη, λέω, ο Σδάγκη. Και δεν μίλησα και για το χάσμα μεταξύ των φίλων, για την Ιρλανδία. Η Κεντρική Τράπεζα έχει μια θετική εκτίμηση για τη σημαντική πρόοδο που πέτυχε η Ιρλανδική κυβέρνηση σε πολύ δύσκολες συνθήκες και αντιμετωπίσαμε επίσης και τις ανησυχίες σε σχέση με τις θυσίες που έχουν γίνει στην Ιρλανδία που ήταν πραγματικά πολύ έντονες. Υπάρχει τώρα αυτό το ειδικό θέμα το οποίο αναφέρατε, το οποίο είναι υποσυζήτηση και ήταν υποσυζήτηση του τελευταίους μήνες. Είναι η προσπάθεια όλων των μερών να βρουν μια λύση για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να, να μην ξεχάσουμε όμως ότι η Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κάνει νομισματική χρηματοδότηση και να αντικαταστήσει αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέρη για τα θέματα αυτά. Αυτό ισχύει και για την Ιρλανδία αλλά και για όλε τι άλλε περιπτώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να θεωρήσει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να υποκαταστήσει κυβερνητικέ δράσει ή κυβερνητική αδράνεια με το να τυπώσει απλώ χρήματα. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μα είναι επίση πολύ νο... απλό να θεωρεί κανείς ότι ένα μικρό κράτο μπορεί να φέρει όλο το φορτίο αυτό. Το φορτίο αυτό είναι τεράστιο. Μιλάμε το 20%, του 120% του ΑΕΠ μας όταν κοινωνικοποιήσαμε το τραπεζικό χρέος. Πρέπει να υπάρξει κάποια κίνηση για τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη έχει πράξει πολλά για τα θέματα αυτά ο κύριο και συνεργάζεται με την Ιρλανδική κυβέρνηση για να μπορέσουν να εξερευνηθούν λύσει. Θα πρέπει όμω να έχουμε στο μυαλό μα ότι όλοι από εμά έχουμε τι δικέ μα ευθύνε και πρέπει να δράσουμε μέσα στα πλαίσια των εντολών μα. Για το θέμα του φύλου. Είπατε ότι εμείς έχουμε την δυνατότητα να διορίσουμε όποιο φύλλο προτιμάμε στο επόμενό μας εποπτικό συμβούλιο. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι αυτό βέβαια εξαρτάται από την τελική νομοθετική ρύθμιση. Όπως σας είπα προηγουμένως, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε στο μυαλό μας και θέλουμε να βρούμε μια πραγματικά, ε, πραγματική ε, λύση για το θέμα αυτό και όχι απλώς φραστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Right, thank you. Thank you very much for that. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, λίγα λεπτά διακοπή. Πριν ε, επανέλθετε με την άλλη σας ιδιότητα. Ο Μάριο μας είπε ότι δεν χάνετε την εποπτεία, είναι σαν να κερδίζετε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αργότερα θα πάμε και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και... Ε, θα επανέλθουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά. Να επαναλάβουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Πρωτού χάσουμε και άλλο χρόνο. Ε, καθίστε παρακαλώ. Θα έχουμε τώρα την ε, παρουσίαση από τον Μάριο για 10 ακόμα λεπτά, ο οποίος τώρα αναλαμβάνει υπό την ιδιότητά του ως ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ίσως υπάρχει μια κάποια επικάλυψη με την προηγούμενη συζήτηση, αλλά τώρα περνάμε στον νομισματικό διάλογο και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα που σας ενδιαφέρει. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Με χαρά σας ξαναβλέπω στο Κοινοβούλιο και με χαρά συναντώ την Επιτροπή σας για την τακτική ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρει σημαντικές αποφάσεις πρόσφατα για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στον τομέα των κρατικών ομολόγων. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε κατά από συγκεκριμένε συνθήκες αυτό το οποίο ονομάζουμε OMTs, οριστικές νομισματικές συναλλαγές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιτρέψει να υπάρξει ένα πλαίσιο αποφυγής καταστροφικών σεναρίων που θα απειλήσουν τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη ευρώ. Η ανακοίνωση την οποία κάναμε για τις οριστικές νομισματικές συναλλαγές βοήθησε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα θα γεφυρώσουν την κατάσταση, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ξεκάθαρη κατεύθυνση. Αυτό για να γίνει χρειάζεται τρεις βασικές διαδικασίες. Πρώτον, μια πλήρη εφαρμογή της δημοσιονομικής αποκατάστασης και των διαφορετικών αλλαγών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεύτερον πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και τρίτον την ολοκλήρωση μιας πραγματικής και γνήσιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Η δημιουργία ενός ενιαίου ελεγκτικού μηχανισμού ή μηχανισμού εποπτείας είναι κομβικό σημείο στις διαδικασίες αυτές. Σήμερα θα επανεξετάσω τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις από το μήνα Ιούλιο και μετά θα εξηγήσω σε επίπεδο λεπτομέρειας την λογική και τους τρόπους που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις οριστικές αυτές νομισματικές συναλλαγές και θα σας παρουσιάσω και τα τέσσερα κεντρικά σημεία της νομισματικής ένωσης και της ένωσης των χρηματαγορών. Μετά από την τελευταία μας συνάντηση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, δεν ε, άλλαξε τα βασικά της επιτόκια. Το βασικό επιτόκιο είναι 0,75% το λεγόμενο αναχρηματοδότησης. Το επιτόκιο καταθέσεων είναι στο 0% και ε, η οριακή διευκόλυνση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1,50%. Η οικονομική δραστηριότητα συρρυκνώθηκε στο δεύτερο τέταρτο του 2012 προοπτικά εμείς προβλέπουμε ε, ασθενείς οικονομικές δραστηριότητες βαχυπρόθεσμα και μια πάρα πολύ σταδιακή ανάκαμψη μετά από αυτό το τέλος του χρόνου. Οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις αυτές ε, μειούνται. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τις εντάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή κυριαρχούν σε πολλές χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο μέσο όρο του πληθωρισμού ήταν 2,7% το Σεπτέμβριο στη ζώνη ευρώ, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει και τους έμεσους φόρους και τις υψηλότατες τιμές ενέργειας. Θα πρέπει να μειωθεί ίσω και κάτω από το 2% κατά τη διάρκεια του 2013. Η πίεση προς τις τιμές θα παραμείνει χαμηλή, μιας και υπάρχουν χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάκαμψης, και ε, θα έλεγα υπάρχουν και κάποιες πρόοπτικες εδώ και αρκετό καιρό για μακροπρόθεσμες πληθωριστικές τάσεις. Οι κίνδυνοι λοιπόν είναι αρκετά μοιρασμένοι. Η νομισματική ανάλυση μας ε, περιγράφει μια εικόνα θα έλεγε η οποία είναι συμβατή με τη σταθερότητα των τιμών. Ο ρυθμός νομισματικής ανάκαμψης είναι σχετικά χαμηλός. Ε, θα έλεγα και η δανειοδοτική δυναμική είναι και αυτή χαμηλή λόγω ακριβώς της χαμηλής ζήτησης αλλά και της ε, ε, περιοριστικής σε αυτή τη φάση προσφοράς απιστώσεων σε ορισμένες χώρες. Να σας εξηγήσω τώρα την απόφαση που πήραμε το Σεπτέμβριο σχετικά με τις οριστικές νομισματικές συναλλαγές. Οι επιπτώσεις σε χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες ε, παλαιών μειώσεων στις, στις ζώνες, στη ζώνη ευρώ προκάλεσαν διαφορετικού τύπου ε, αλλαγές στις διάφορες χώρες. Δηλαδή σε ορισμένες ε, χώρες όταν μειώσαμε εμείς τα επιτόκια, τα επιτόκια τα οποία χρησιμοποίησαν τα τραπεζικά του συστήματα είτε δεν μειώθηκαν καθόλου είτε μειώθηκαν πολύ λίγο. Ενώ σε άλλες χώρες ε, τα επιτόκια τα μειωμένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πέρασαν αυτόματα. Ένας λόγος για αυτή την διαφορά είναι ότι το κόστος ε, πρόσβασης σε πίστοση από τις, από τις τράπεζες της επιχειρήσης συνδέεται άμεσα από το κόστος δανειοδότησης των ιδίων των τραπεζών μεταξύ τους. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτούς τους φόβους θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε γιατί επηρεάζονται ασυμμετρικά θα έλεγα οι διάφορες χώρες και οι διάφορες τράπεζες στην ευρωπαϊκή ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι δύο επιχειρήσεις οι οποίες είναι ταυτόσιμες, έχουν την ίδια αξία και σε επίπεδο δανειοδότησης, ε, μπορεί να δανειστούν με διαφορετικά ποσοστά μόνο και μόνο επειδή είναι σε δύο διαφορετικές χώρες. Πρόκειται για μια στρέβλωση στο κόστος της χρηματοδότησης που παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία των πιστοτικών αγορών και την μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Αυτή ακριβώς η στρέβλωση κρατάει ορισμένες χώρες τις οποίες ε, έχω, σε μια κατάσταση την οποία έχω ε, θα έλεγα ονομάσει και στο παρελθόν κατάσταση κακής ισορροπίας. Και αυτή ακριβώς τη στρέβλωση πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της εντολής μας. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τις δυσκολίες μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και να διατηρήσουμε τον ενιαίο χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής, εμείς προσπαθήσαμε, αποφασίσαμε μάλλον να περάσουμε στα λεγόμενα OMT, δηλαδή στις οριστικές νομισματικές συναλλαγές για να αποφύγουμε καταστροφικά σενάρια που θα απειλούσαν τη σταθερότητα των τιμών. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μεταδίδεται με πιο σωστό και ισότιμο τρόπο στην πραγματική οικονομία στο σύνολο της ζώνης ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει με τα OMT εφόσον οι χώρες και όσο καιρό οι χώρες συμφωνούν με τις προϋποθέσεις τις αυστηρές και τις ουσιαστικές ε, που έχουν καθοριστεί μέσω του Ευρωπαϊκού ε, Μηχανισμού Σταθερότητας και του ε, Ευρωπαϊκού Σταθεροποιητικού Μηχανισμού. Η ερεσιμότητα διατηρεί, θα έλεγα, την βασική μας εντολή και δεν θα αντικαταστήσει την έλλειψη δράσης στον τομέα των δημοσιονομικών. Η αιρεσιμότητα ταυτόχρονα διατηρεί τα κίνητρα για τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν με τις οικονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις. Και μόνο εφόσον εκπληρούνται οι όροι αυτή της αιρεσιμότητας θα μπορέσουν τα OMT, αυτές οι τελικές ή οριστικές αν θέλετε νομισματικές συναλλαγές, να οδηγήσουν την οικονομία σε μια καλή ισορροπία υπάρχει δυνατότητα, θα έλεγα, να θεωρήσουμε ότι αυτές οι οριστικές συναλλαγές είναι απεριόριστες εκ των προτέρων. Αλλά υπάρχουν πάντα ορισμένες προϋποθέσεις. Η έξοδος από τα OMT μπορεί να γίνει όταν οι στόχοι τους έχουν πλέον ολοκληρωθεί ή όταν υπάρχει αποτυχία, θα έλεγα, στο πρόγραμμα. Τα OMT δεν θα υπάρχουν, δεν θα ε, δίδονται όταν ένα πρόγραμμα είναι σε περίοδο αξιολόγησης και θα συνεχίζονται εφόσον έχει διασφαλιστεί, θα έλεγα, έχουν διασφαλιστεί οι συνθήκες οι οποίες προαπαιτούνται. Σύμφωνα πάντα και με τη συνθήκη που απαγορεύει την χρηματοδοτική ε, άμεση χρηματοδότηση, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, θα παρεμβαίνει αυστηρά σε, σε δευτερογενείς αγορές και όχι σε κυβερνήσεις αλλά σε ιδιώτες επενδυτές. Σύμφωνα πάντα με τις ε, παραδοσιακές θα έλεγα μορφές δραστηριοποίησή μας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούμε με τον ίδιο τρόπο με άλλους ιδιώτες πιστωτές σε σχέση με τα ομόλογα τα οποία αγοράζουμε στα πλαίσια των OMT. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι απολύτως διαφανής. Εμείς σε αιτήσια βάση θα αναφερόμεθα στο τι έχουμε στην διακατοχή μας και σε μηνιαία βάση για τη διάρκεια των, του ενεργητικού μας αναχώρα. Να περάσω τώρα στο άλλο θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει σήμερα, το θέμα της χρηματοπιστωτικής ένωσης, αν θέλετε. Εμείς δεχόμαστε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Είναι κάτι το οποίο είναι συμβατό με την απόφαση της συνάντησης κορυφής της 29ης Ιουνίου. Εμεί προσδοκούμε να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό. Είμαι πεπισμένο ότι η εξαιρετική συνεργασία την οποία μέχρι τώρα έχουμε πετύχει θα συνεχιστεί και στο μέλλον στον τομέα της χρηματοπιστωτική εποπτείας. Να συγκεντρώσω την προσοχή μου τώρα, αν μου επιτρέψετε, σε τρία θέματα, τα οποία είναι κομβικά για την δημιουργία ενός νέου διακανονιστικού εποπτικού πλαισίου στη ζώνη ευρώ. Πρώτον, η αρχή του διαχωρισμού ανάμεσα στην νομισματική πολιτική και στην χρηματοπιστωτική εποπτεία. Δεύτερον, η πιθανότητα συμμετοχής χωρών μελών εκτός ζώνης ευρώ. Και τρίτον, το λεγόμενο πλαίσιο λογοδοσίας. Στο πρώτο θέμα του διαχωρισμού της νομισματικής πολιτικής και των ελεγκτικών λειτουργιών, νομίζω ότι έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο. Πολλές κεντρικές τράπεζες στον κόσμο μεταξύ των οποίων και η μεγάλη πλειοψηφία των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο ευρωσύστημα, συνδυάζουν τις νομισματικές αποστολές με τις ελεγκτικές. Θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις έτσι ώστε η νομισματική πολιτική να μην επηρεαστεί αρνητικά από τον ελεγκτικό ρόλο και αυτό ισχύει σε πολλές χώρες ήδη. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε εμείς να καταλήξουμε σε κατάλληλες ρυθμίσεις και στη ζώνη ευρώ ε, εκμεταλλευόμενοι τις δικές τους εμπειρίες, τις εμπειρίες των επιμέρους χωρών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια σωστή βάση λοιπόν μέσω του ελεγκτικού μηχανισμού ο οποίος θα κάνει τις τακτικές ε, ε, εποπτικές δραστηριότητες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μπορέσουμε να αποφύγουμε κάποιες συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στις δύο λειτουργίες. Ταυτόχρονα Εξετάζουμε τώρα τις εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες θα ξεχωρίσουν τις διοικητικές δραστηριότητες που ασχολούνται με τις δύο αποστολές. Το δεύτερο κομβικό αν θέλετε πλαίσιο για τον εποπτικό μηχανισμό είναι η δυνατότητα συμμετοχής χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη και που θέλουν να πάρουν μέρος στο SSM. Καταρχάς, ας θυμηθούμε γιατί δημιουργούμε την χρηματοπιστωτική αυτή ένωση, λόγω ακριβώς το τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη σήμερα. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να σπάσουμε το φαύλο κύκλο ανάμεσα στο δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, οι συνέπειες ε, του οποίου αυτού φαύλου κύκλου είναι πάρα πολύ θα έλεγα, ε, είναι οξύτατες ε, στην νομισματική ένωση. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε το SSM. Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε την ένωση αυτή, την χρηματοπιστωτική, ενισχύοντας την ενία αγορά και το ενιαίο νόμισμα και ενιαία αγορά είναι δύο πυλώνες ανάπτυξης και ευημερία στην Ευρώπη. Και οι δύο αυτοί πυλώνες θα πρέπει να διατηρηθούν και να βελτιωθούν. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί πολύ θετική τη δυνατότητα συμμετοχής χωρών εκτός ζώνης ευρώ στο SSM. Η συμμετοχή επιπλέον μελών θα δημιουργήσει, θα έλεγα, μια καλύτερη και ισχυρότερη όθηση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Πέραν τούτου, και για ένα όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, των οποίων οι νομικές, θα έλεγα, αρμοδιότητες και τα φόρα λήψης απόφασης είναι περιορισμένα στη ζώνη ευρώ, το να επιβάλλει κάποιες υποχρεώσεις και να δίδει αντίστοιχα δικαιώματα σε χώρες εκτός ζώνης ευρώ θέτει ορισμένα νομικά θέματα. Οι νομικέ μα υπηρεσίε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο εξετάζουν προσεκτικά τι πιθανέ τροποποίησει στη συμμετοχή χωρών εκτό ζώνη ευρώ στα πλαίσια των νομικών περιορισμών ε, του κανονισμού μα. Το τρίτο θέμα λοιπόν για το ελεγκτικό πλαίσιο είναι αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πώς θα είναι υπόλογη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις εποπτικές της δραστηριότητες προς τους πολίτες της Ευρώπης και τους ε, ε, βουλευτές τους οποίους ο ευρωπαϊκός λαός εκλέγει. Ε, η ανεξαρτησία αυτής της εποπτικής θα έλεγα δραστηριότητα είναι σημαντική αλλά πρέπει να είμαστε υπόλογοι και το ένα και το άλλο λαμβάνοντας υπόψη της φύσης, τη φύση της εποπτείας και την ανάγκη της συνεργασίας με άλλες αρχές, εκεί όπου θα υπάρχει και δημοσιονομικό κόστος, είναι σαφές ότι ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι ισχυροί μηχανισμοί ε, ε, που θα καθορίζουν ακριβώς το υπόλογο της τράπεζας αλλά και θα νομιμοποιούν το υψηλό ποσοστό ανεξαρτησίας. Θα πρέπει να είμαι το SSM υπεύθυνο και υπόλογο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα πρέπει να δούμε τώρα και πώς θα, πότε θα ξεκινήσουμε ανεξαρτήτως ε, του χρονοδιαγράμματος ε, για την άσκηση των ε, εποπτικών αρμοδιοτήτων, νομίζω ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου του 2013. Αυτό θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε τις προπαρασκευαστικές εργασίες το ταχύτερο δυνατόν. Έχω εξετάσει ήδη τα βασικά χαρακτηριστικά του SSM, αλλά η Ένωση η Χρηματοπιστωτική θα είναι ατελής εάν δεν υπάρξει σημαντική πρόοδος και προς ένα θα έλεγα κοινό καθεστώς επίλυσης διαφορών. Η έλλειψη ενός τέτοιου καθεστώτος έχει αυξήσει το κόστος των αποτυχιών των τραπεζών για τον φορολογούμενο και έχει περιπλέξει τα πράγματα ιδιαίτερα σε διαμεθοριακά φαινόμενα αποτυχίας. Θα πρέπει λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Αρχή ε, να λειτουργήσει σωστά για να ελέγξει κρίσεις με σωστό, αποτελεσματικό και τακτό τρόπο. Για να κλείσω, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωζώνη έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου για να βελτιώσει και να εξηγιάνει τα θεμελιά της. Νομίζω ότι τον Οκτώβριο και αργότερα τον Δεκέμβριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα επιβεβαιώσουν την πορεία προς το αναπόδραστο του ευρώ, συμφωνώντας ε, σε ένα όραμα μακροπρόθεσμο για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η διαδικασία αυτή δεν έχει επηρεάσει ξεκάθαρα την καθημερινότητα του πολίτη στις χώρες οι οποίες υποφέρουν περισσότερο από την κρίση. Συνειδητοποιώ τις δυσκολίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η παρούσα κατάσταση για πάρα πολλούς πολίτες ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τη θέση εργασίας τους ή είναι σε κίνδυνο η θέση εργασίας τους. Οι διαδικασίες ρύθμισης προς ε, βιώσιμα δημοσιονομικά και μια ανταγωνιστική οικονομία είναι κάτι το οποίο θα είναι οδυνηρό, βραχυπρόθεσμα, πολιτικά, οικονομικά και ανθρώπινα. Όμως οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες, είναι διορθώσεις αυτές οι μεταρρυθμίσεις που θα επαναφέρουν τις χώρες ε, ε, στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη και θα συνεισφέρουν στην κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της σωστής φορολόγησης και μέσω της μείωσης της σημασίας των επενδεδημένων συμφερόντων. Είμαι πεπισμένος ότι ε, από την κρίση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει με πιο ισχυρές και καλύτερα λειτουργούσες οικονομίες προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρώπης. Um, Ωραία. Τι θα κάνω τώρα. Πάλι ομαδικά οι ερωτήσεις, ανά κερδίζουμε έτσι κάπως χρόνο. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν και επικαλύψεις. Συνεπώς, οι πρώτοι τρεις είναι Πάλτς, Φερέιρα και Γκουλάρ. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω κάποια ερωτήματα στον κύριο Τράκη για το θέμα της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές μηχανισμ... αγορές. Μιλήσατε για ένα μηχανισμό εποπτείας ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και την Κεντρική Τράπεζα. Ναι, ναι, μια στιγμή χρειαζόμαστε να βάλουμε τα ακουστικά μας, λέει η Σάρων. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω ερωτήματα για την Ένωση, χρηματο... στην Χρηματοπιστωτική Ένωση υπήρξε αυτή η απόφαση για ένα εποπτικό μηχανισμό με συμπερίληψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τραπεζάς. Have to put it <laughs> Ξαναμηδενίστε όμως το χρονόμετρο, λέει ο κύριος Μπάλτς. Είπαμε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έδωσαν μια εντολή για τη δημιουργία ενός εποπτικού μηχανισμού, ο οποίος να συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά, η φήμη και η εμπειρογνωμοσύνη της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το κάνει αυτό εύλογο. Εγώ φυσικά έρχομαι από τη Γερμανία και επομένως εκτιμώ ιδιαίτερα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι γίνεται όμως <clears throat> αν δεν λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός καταρχήν, ο εποπτικός μηχανισμός υπάρχουν κίνδυνοι να πληγεί και η φήμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι πράγματι προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εξασφαλίσει ότι θα συμμετέχει περισσότερο στους ήδη υπάρχοντες φορείς εποπτείας. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Για τη συμμετοχή των μη, των χωρών που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος Υπάρχει κίνδυνος να υπάρχει και κάποιο ρήγμα μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω εδώ ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο μπορεί να έχει συντριπτικό χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες είναι στο δρόμο στην ένταξη της ε, ζώνης του ευρώ. Μήπως θα ήταν καλύτερο για τον εποπτικό μηχανισμό, αντί να έχουμε ένα μηχανισμό ε, opt-in, να έχουμε μηχανισμό opt-out. Όχι αυτό ε, αποδοχή αλλά μηχανισμό αυτοεξαίρεσης, opt-out. Να ξέρουμε λοιπόν ποιες χώρες δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτόν τον φορέα, τον εποπτικό και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό μέσα στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της δομές της. Η Ελίζα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις αποφάσεις που πήρε, ιδίως για τις οριστικές νομισματικές πράξεις ή συναλλαγές, γιατί αυτό ήταν ένα μήνυμα το οποίο οδήγησε σε ανακούφιση και έδωσε εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ντράγκη να μου πει αν έχει κάποιο όραμα για το μέλλον σε σχέση με αυτές τις πράξεις, αν είναι απλώς μια αν βλέπει ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να εξασφαλίσει την διασφάλιση του κρατικού χρέους και την αναζωγόνηση της αγοράς, αν μονάχα μια ψηφίδα σε ένα ευρύτερο σχέδιο. Επίσης, τώρα στο θέμα της αιρεσιμότητος, και εδώ συνδέεται με το προηγούμενο ερώτημά μου. Όταν υπάρχει η επιβολή μιας αιρεσιμότητας στις χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις συναλλαγές, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η τοποθέτηση, ποια είναι η θέση της Κεντρικής Τράπεζας. Φυσικά χρειάζεται να υπάρξει μια οικονομική ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Όταν όμως τηρούνται κάποιες ε, επιβολές που οδηγούν σε μια οικονομία η οποία συρρυκνώνεται και αυτό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε, αναρωτιέμαι αν η Κεντρική Τράπεζα θέλει να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει την ποιότητα των ε, συστάσεών της, ιδίως αν είναι τμήμα μιας τρόικας. Θέλω λοιπόν να δω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει να προκύψει και κάποια προοπτική ανάπτυξης αυτή τη στιγμή από αυτή την αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να δω από πού μπορεί να έρθει μια δυναμική ανάπτυξη, μια αναζωγόνηση της ζήτησης. Όταν οι χώρες αυτές λοιπόν είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν πολιτικές λιτότητας, είτε έχουν πλεόνασμα είτε έχουν έλλειμμα, <clears throat> ελείπει η πηγή της ζήτησης που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Επίσης δεν υπάρχει η κατανομή των βαρών για τα θέματα επίλυσης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κατεπήγον να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους θα μπορέσουν επί της ίδιας βάσης να συμμετέχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο, ταμείο, ε, στο μηχανισμό επίλυσης. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να παραμείνει αποσυνδεδεμένος από το μηχανισμό εγγύησης καταθέσεων. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Γκούλαρ. Δεν θα ρωτήσω τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με την σύνθεση του Ταμείου για τον Έλεγχο για την εποπτεία θα μου δώσετε τα στοιχεία του θαυμάσιου προσωπικού που έχετε στην τράπεζά σας λέγοντας ότι σε νομικό επίπεδο δεν έχετε καμία σχέση με όλα αυτά, ότι είναι αυτό μια απόφαση του Συμβουλίου και ίσως εν καιρό θα υπάρξει και μια γυναίκα στο Εποπτικό Συμβούλιο. Και τώρα περνάω στα Ιταλικά. Θα ήθελα να πω στο Μάριο, όχι στον Πρόεδρο, αλλά στο Μάριο, στον άνθρωπο που είναι λογικός πώς βλέπει να πάμε τα επόμενα 7 χρόνια. Είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνο για ένα θεσμικό όργανο το οποίο ζητάει από όλη την Ευρώπη αναδιάρθρωση, εξυγχρονισμό, περισσότερες γυναίκες στη δουλειά, αλλά είναι πάντα αφεντικό σε εισαγωγικά ενός οργάνου το οποίο λειτουργεί με κανόνες του παρελθόντος. Έχει μόνο άνδρες Χθες ακούστηκαν πολλοί οικονομολόγοι στο Vox EU να ζητούν λιγότερες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Πώς πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να αξιολογήσει κανείς το υπόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Πιστοντικής Τραπεζικής Ένωσης εάν το Συμβούλιο δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη αυτά τα οποία λέει το Κοινοβούλιο, τα αγνοεί συστηματικά. Μιλάτε εξαιρετικά Ιταλικά, ανταποδίδει ο κύριος Ντράγκη. Για το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε τη σχέση μεταξύ του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και των υπαρχόντων δομών εποπτείας. Νομίζω το είπα και στην αρχή. Ήταν η πρώτη μου ίσως δημόσια δήλωση μετά από την πρόταση της Κομισιόν, μετά από το Συμβούλιο του Ιουνίου που ξεκίνησε αυτή την αντιμετώπιση για το συστημικό έλεγχο, τον εποπτικό μηχανισμό. Είχαμε εθνικούς εποπτικούς φορείς που στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι σε όλες, είχαν δείξει ικανότητα αντιμετώπισης, είχαν την γνώση της χώρας τους, ξέραν την τραπεζική ιστορία της χώρας τους και είχαν πολύ ικανό προσωπικό. Θα ήταν αδιανόητο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προσπαθήσει να τους αντικαταστήσει. Αλλά έκτοτε εμείς έχουμε συνεργαστεί μαζί τους σε, μεγάλο ενεργό, σε πολύ ενεργό επίπεδο και αυτό το οποίο τους είπα στην τελευταία συνάντηση που είχαμε είναι ότι εμείς είμαστε αναπόσπαστο τμήμα του ίδιου εγχειρήματο. Δεν είναι ότι θέλουμε να διασπάσουμε την εποπτεία σε δύο χώρου. Όχι. Θα αποφασίσουμε από κοινού, γιατί και αυτοί θα εκπροσωπούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο. Θα παίρνουν κοινέ αποφάσεις όλοι αυτοί οι φορείς από κοινού. Θα είναι πολύ φυσικό να αποφασίσουμε ποια εγχειρήματα και ποια καθήκοντα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κεντρικά και ποια τοπικά και ποιες τράπεζες θα πρέπει να εποπτεύονται τοπικά και ποιες ε, κεντρικά. Αλλά ακόμα και αν τα καθήκοντα αυτά γίνονται σε κεντρικό επίπεδο, οι εθνικοί επόπτες θα είναι τμήμα τη λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, γιατί υπάρχει μια φυσική τάση να θεωρεί κανεί ότι η εποπτεία μπορεί να γίνεται είτε από τη Φραγκφούρτη είτε από τι Εθνικέ Εποπτικέ Αρχέ. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κοινή η διαδικασία λήψεων αποφάσεων σε σχέση με την εποπτεία. Είναι προφανέ ότι θα υπάρχουν και κάποιοι, κάποιοι, κάποια καθήκοντα όπω οι επιθεωρήσει που θα είναι πιο φυσιολογικό να γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Σε άλλε επιπτώσει θα είναι πιο λογικό να γίνονται σε κεντρικό επίπεδο. Πάντα όμω θα γίνεται κάτι τέτοιο με τη συμμετοχή των εθνικών φορέων εποπτικού χαρακτήρα. Για το δεύτερο ερώτημά σας για τις χώρες που δεν είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ και τη συμμετοχή τους. Η θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εδώ είναι απόλυτα ανοιχτή. Τα, οι χώρες που δεν είναι μέλη της ε, ζώνης του ευρώ προσκαλούνται να είναι τμήμα αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, κατά την άποψή μα, θα πρέπει να έχουν ακριβώ τα ίδια δικαιώματα όπω οι χώρε που είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ. Εμεί πρέπει να συμβιβάσουμε κάτι τέτοιο με ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν κάνει ιδιαίτερα προφανές πώς θα συμμετάσχουν αυτές οι χώρες. Όλοι μας εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση όμως με την ελπίδα να βρούμε μια λύση. για τις ε, οριστικές ε, νομισματικές συναλλαγές. Όπως σας είπα, με τον τρόπο αυτό έχουμε ένα πραγματικό ανάχωμα το οποίο αποτρέπει τους λεγόμενους κινδύνους ουράς από την περιοχή του ευρώ εφόσον τηρηθούν ορισμένε προϋποθέσεις. Κατά κάποιο τρόπο το ερώτημά σας, η απάντηση μάλλον προς το ερώτημά σας είναι η εξή ξεκινώντας από το τέλος του ερωτήματά σας. Από πού θα προέλθει η οικονομική μεγέθυνση. Μπορεί να έρθει από μια δημοσιονομική πολιτική, δεν μπορεί να έρθει μάλλον από τις δημοσιονομικές πολιτικές, συγγνώμη, από πού μπορεί να προέλθει επομένω. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να προέλθει από το χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων. Αλλά το χαμηλό επί επίπεδο των επιτοκίων δεν ε, μεταφράζεται σε ένα, σε ένα χαμηλό επίπεδο επιτοκίων δανεισμού που είναι το σημαντικό για την πραγματική οικονομία και ο λόγος που δεν γίνεται κάτι τέτοιο είναι ο κατακαιρματισμός της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας λοιπόν η μεγαλύτερη συνεισφορά στην ανάπτυξη είναι να ξεπεράσουμε την τωρινή κατάσταση κατακαιρματισμού στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Όταν λέμε να επιδιορθώσουμε τους μηχανισμούς μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής σημαίνει ότι θα επιδιορθώσουμε τους μηχανισμούς ώστε να ξαναρχίσει ο δανεισμός να μην είναι βουλωμένη η διάβλη δανεισμού όπως είναι αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει τόσο μεγάλη ψαλίδα στα βραχυπρόθεσμα πρόθεσμα επιτόκια κτλ. Φυσικά η η οικονομική μεγέθυνση θα πρέπει να γίνει και με την εξάλληψη των οικονομικών ακαμψιών και την διαρθρωτική αλλαγή. Εμείς προσπαθούμε να άρουμε ένα από τους λόγους της, ε, ε, του κατακαιρματισμού της μη λειτουργίας του νομισματικού μηχανισμού μετάδοσης που είναι η κίνδυνη ουρά, risks, η κίνδυνη να βγει μια χώρα από το ευρώ. Επίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν το τον στρεβλό κύκλο που συνδέει το κρατικό χρέος με το τραπεζικό χρέος. Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο και το σχέδιό μας να έχουμε ένα ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, μία αρχή επίλυσης και όπως είπα εν καιρό μία ενιαία ε, διαδικασία εγγύησης καταθέσεων, Αυτή είναι οι τρεις μηχανισμοί με τους οποίους θα σπάσουμε αυτό το φαυλοκύκλο σύνδεση δημοσίου χρέους και τραπεζών. Αλλά η μεγαλύτερη συνεισφορά προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνει μονάχα με το να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της, ε, του κατακαιρματισμού της χρηματοπιστωτικής αγοράς που έχει πλήξει την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία τρία χρόνια για την αιρεσιμότητα που αναφερθήκατε. Μπορώ να πω ότι εμείς δεν επιβάλλουμε προϋποθέσεις. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία κάνει κάτι τέτοιο. Ζητούμε ως μία απαραίτητη αλλά ως ικανή συνθήκη οι χώρες να προσυπογράψουν ένα πρόγραμμα στα πλαίσια του e F και του ESM και θα ζητήσουμε και την αρρωγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την αξιολόγηση της ερεσιμότητας. Γιατί το πράγμα αυτό, διότι είμαστε πεπισμένοι ότι η νομισματική μας πολιτική ακόμα και αν έχει στοιχεία έκτακτα όπως είναι οι δράσει οριστικών νομισματικών πράξεων, θα επηρεαστούν αν οι εμπλεκόμενες χώρες δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Όπως έχω πει και σε άλλες περιφτάσεις, ξεκινάμε από χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός ισορροπίας. Δηλαδή έχουμε ε, προσδοκίες οι οποίες οδηγούν πάντα σε αρνητικά σενάρια, όσο και να κάνει πρόοδο μια χώρα. Επομένως, είναι υποχρεωμένη να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αρκεί αυτό, όχι. Γιατί δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε πώς οι χώρες αυτές βρέθηκαν εκτός ισορροπίας. Βρεθήκαν εκτός ισορροπίας διότι ακολούθησαν λανθασμένες οικονομικές πολιτικές ή αδράνησαν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες πολιτικές για 10 χρόνια ενώ ο κόσμος γύρω τους άλλαζε. Είναι σαν τα δύο πόδια. Χρειάζεται κανείς δύο πόδια για να περπατάει. Και αυτή είναι η λογική της αιρεσιμότητας. Το τρίτο ερώτημα είναι η κατανομή του βάρους. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα κύρια προβλήματα για το σχεδιασμό του Ταμείου Επίλυσης. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα, αλλά θα πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε, γιατί το Ταμείο Επίλυσης αυτό καθεαυτού δεν θα πρέπει να είναι μεγάλο, δεν είναι ένα ταμείο διάσωσης, είναι ένα ταμείο επίλυσης. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την διαδικασία διάσπασης τραπεζών που έχουν επιληθεί θα πρέπει να χρηματοδοτήσει στο διάστημα όταν αποφασίζει κανείς ποια κομμάτια της τράπεζας θα διατηρηθούν εν ζωή και ποια θα διαλυθούν. Ποιοι θα είναι οι πιστωτές μιας τράπεζας οι οποίοι θα πρέπει να αποζημιωθούν και ποιοι όχι και σε ποιο βαθμό. Επομένως, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το νομικό πλαίσιο και το νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία αυτού του Ταμείου Επίλυσης, ώστε να μπορέσουμε βάσει αυτού να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένας μονάχα μηχανισμός σε νομικό επίπεδο για την επίλυση τραπεζών σε όλο τον χώρο του ευρώ. Το τέταρτο ερώτημα που θέσατε αφορά εμένα τον ίδιο αν θέλετε. Ε, κατά 100% εγώ υποστηρίζω τον εξυγχρονισμό. Το ξέρετε και από τις προηγούμενες εμπειρίες μου. Προσπαθώ ουσιαστικά να αντιμετωπίσω τον τρόπο με τον οποίο έχουν λειτουργήσει οι θεσμοί και έχω μεγάλη εκτίμηση και για σας και για το προσωπικό το οποίο έχω υπό τις εντολές μου. Όλοι μας όμως μπορούμε να βελτιωθούμε με πολλούς τρόπους και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο αναφέρατε. Το θέμα του φύλου. Και σας λέω και πάλι δεν υπάρχουν διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εναντίον των γυναικών. Τούτου λεχθέντος όμως ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως και όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς μπορούν να κάνουν πολλά για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και εγώ σας υπόσχομαι να είμαι πάρα πολύ ενεργός στο θέμα αυτό. Μα όταν έχετε 23 άνδρες οι οποίοι αποφασίζουν αυτό είναι διάκριση. Σταματήστε να αποστρέφετε το βλέμμα σας από την πραγματικότητα. Είναι πράγματι μια διάκριση κάπου έχουν πάει τα πράγματα στραβά. Μα εμείς δεν διαλέγουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λέω ο πρόεδρος Τράκη. Είναι οι εθνικές αρχές που μας στέλνουν τα μέλη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ ρωτούσα, ζητούσα από τον Μάριο Τράγκη να κάνει προσωπικά κάποια σχόλια. Ναι, ναι, μπορείτε να βασιστείτε στη δική μου προσωπική ε, αντιμετώπιση. Όπως έλεγα προηγουμένως στην ακρόαση για το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δείτε τα τελευταία δέκα χρόνια, μιλάμε για μια χρηματοπιστωτική κρίση. Τα τελευταία δέκα χρόνια όλες αυτές οι κρίσεις έχουν αντιμετωπιστεί από άνδρες. Είναι καιρός λοιπόν να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Ευχαριστώ. Ωραία. Την κρίση την οφείλουμε στους άντρες. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα, Θέλω να επενθυμίσω στο Μάριο ότι ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως πολύ σημαντική να φροντίσει, να βοηθήσει και επηρεάζοντας τις άλλες κεντρικές τράπεζες να έχουν μια στρατηγική υπέρ της παρουσίας των γυναικών έτσι ώστε να μην ε, είναι πάντα ανδροκρατούμενοι. Πάντα ήταν ε, ανδροκρατούμενες οι διάφορες ε, εθνικές κεντρικές τράπεζες. Εμείς έχουμε πιέσει εδώ και καιρό να αλλάξει αυτό. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Α, πρέπει να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Ρόζα Μπίντιγκ που είναι εδώ από την Πούντεστακ. Ζαμπόλ, διαδικαστικό. Ναι, θέλω να αποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία, μια που το θέμα φαίνεται να είναι πιο σημαντικό όσον αφορά και την Τραπεζική Ένωση. Θέλω να ξέρω πότε θα οριστεί το νέο μέλος ε, της διεύθυνσης της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν ε, δεν απατάμε, από εσά εξαρτάται. Να μένα όχι, λέει ο κύριο Γκοντζές. Εμεί, λέει πρόεδρο, είμαστε στα χέρια του Συμβουλίου. Καλωσορίζω πίσω εδώ και μια αντιπροσωπεία Αμερικανούς από το Marshall Fund των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Πού είσαστε? Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Και τώρα <clears throat> επιστρέφουμε στις εργασίες μας. Α, όχι, κάτι άλλο, ναι. όχι. Ντέρκ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, μιλάμε για τις τράπεζες. Αλλά θέλω να, μιλήσω λίγο, να μιλήσουμε και για τη δικιά σας τη τράπεζα. Μιλάτε για την εποπτεία, για την εμπιστοσύνη. Έχουμε ακόμα δύο χρόνια, αλλά εντωμεταξύ το έχει ανέβει το ποσό από 850 εκατομμύρια σε 1,2 δις. Κάτι το οποίο πληρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Μιλάτε για λιτότητα, αλλά οι ίδιοι δεν ε, επιβάλλεται λιτότητα. Κύριε Ντράγκη, στη Φραγκφούρτη θα κάνετε βέβαια ό,τι μπορείτε, φαντάζομαι. Η πρώτη ερώτησή μου τώρα, είναι μια που συμμετέχουμε στην Τρόικα, είναι ότι για τους Έλληνες, τους Πορτογάλους και τους Ιρλανδούς τους πιέζεται για αυστηρές περικοπές, ε, τεράστιες περικοπές δαπανών. Οι χώρες αυτές όμως πρέπει να συνεισφέρουν συγχρόνως περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν αρκετά για τις δαπάνες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πώς το δικαιολογείται αυτό. Και αν δείτε τη μακέτα του κτηρίου, είναι πραγματικά διάφανο απ' έξω, αλλά από μέσα είναι, υπάρχει διαφάνεια. Και αν ε, για τη δημοσίευση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου θα τα δημοσιεύετε, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για όλους. Συνεχίζουμε. Η Εύα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δικητά, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε κάτι όσον αφορά τις οριστικές νομισματικές συναλλαγές. Στις 6 Σεπτεμβρίου ακούσαμε ότι οι συναλλαγές αυτές θα εφαρμόζονται στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα εξυγίανσης και που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους προς τις αγορές. Αλλά στην τελευταία συνέντευξη τύπου είπατε ότι οι συναλλαγές αυτές ε, θα επιτρέπονται μόνο για χώρες οι οποίες έχουν ε, βρεθεί και πάλι στις ε, αγορές και μπορούν να δανειστούν από τις αγορές. Μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτή την αντίφαση. Τώρα υπό το φως των προεργασιών για μια τραπεζική ένωση, εσείς είπατε ότι πρέπει να διασφαλιστεί διαχωρισμός ανάμεσα στην νομισματική πολιτική και την πολιτική μακροπροληπτικής εποπτείας. Και αναφερθήκατε στην ε, σύγκρουση συμφερόντων και είπατε ότι πρέπει να αποφευθεί. Θέλω να μου διευκρινίσετε περισσότερο τι κίνδυνος υπάρχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή κατά τη γνώμη σας υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων από την αποστολή στην νομισματική πολιτική και την εποπτεία εφόσον δεν υπάρξει τέτοια διάκριση. Και να μας πείτε επίσης τι συνέπειες μπορεί να έχει αν ε, μεταφερθεί αρμοδιότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ένα άλλο συμβούλιο ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα λογοδοτεί. Κατά τη γνώμη σας, οι διατάξεις του άρθρου 130 της συνθήκης εφαρμόζονται στα προνόμια ενός ενδεχομένου μελλοντικού συμβουλίου εποπτών ή από την άλλη, εσείς βλέπετε τη δυνατότητα από τον νομοθέτη να μπορεί δημοκρατικά να ελέγχει περισσότερο σε περίπτωση που περνάνε υποπτικές αρμοδιότητες ε, σε άλλα χέρια. Για παράδειγμα, πώς θα γίνεται ο δημοσιονομικός έλεγχος και έρευνες. Έπειτα, τι, ποιος θα είναι ο διαιτητής, εσείς. Θέλω επίσης να επωφεληθώ από την ευκαιρία που έχω το λόγο για να στηρίξω αυτό που ζήτησαν και άλλοι συνάδελφοι και να πω και εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο φίλων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η σημερινή κατάσταση είναι σκανδαλώδης. Για να μην μιλήσω και για την ανάμειξη του Golden Sachs. Η Μαρίσα Ματέης τώρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ντράγκη σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να επανέλθω στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα προσαρμογής και θα σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι λειτουργούν αυτά τα προγράμματα προσαρμογής και εξυγίανσης. Γιατί είπατε πολλές φορές ότι είπατε ότι είναι προγράμματα τα οποία θα είναι οδυνηρά για τους πολίτες, θα δημιουργούν πολλά προβλήματα και στον χώρο απασχόλησης. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτό αλλά γιατί τα προγράμματα αυτά επιδεινώνουν την ύφεση. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι θετικά αυτά τα προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πλεγμένη σε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία. Εάν η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ε, εξυγίανσης αν θα επαρκέσει. Βλέπετε τι έγινε στην Ελλάδα που υποχρεώθηκε να δεχθεί αυτή τη λιτότητα και τα πράγματα δεν προχωρούν. Πόσα λοιπόν προγράμματα εξυγίανσης θα χρειαστούν. Λέτε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος. Αλλά και πάλι θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι οι δείκτες που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Κεντρικής Τράπεζας για να δει κατά πόσο υπάρχει πράγματι μια πρόοδος όταν μειώνεται συνέχεια η απασχόληση <clears throat> και αυξάνεται και το χρέος και το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Τελικά αξίζει τον κόπο άξιζε τον κόπο να γίνουν όλες αυτές τις θυσίες για, τους, για να, με τα συστήματα, προγράμματα εξυγίανση. Καθυστερούμε λιγάκι, λέει η Πρόεδρος, γιατί τα ερωτήματα ήταν λιγάκι μακροσκελή. Ο κ. Δράγκη, για το κόστος του κτηρίου πρώτα απ' όλα. Ε, αυξάνεται το κόστος για δύο λόγου. Το ένα είναι ο πληθωρισμό που έχει να κάνει με τον οικοδομικό τομέα και τα υλικά που ακριβένουν. 300 εκατομμύρια η διαφορά είναι. Το άλλο τμήμα είναι τα 50 εκατομμύρια που έχουν να κάνουν με τις διάφορες συμβάσεις νομικού χαρακτήρα. Οπότε στα 50 εκατομμύρια μόνο πρέπει να βασίστε τη διαφορά. Για τα πρακτικά σίγουρα θα ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Αλλά εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει διαφάνεια επειδή δεν υπάρχουν τα πρακτικά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα όργανο με διαφάνεια και αυτό φαίνεται από τις ε, δημοσιεύσεις, τις ομιλίες, τις, ε, τα δελτία, τις συνεντεύξεις τύπου, τα ανακοινοθέντα. Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κεντρική τράπεζα στον κόσμο πρέπει να δημοσιεύονται τα πρακτικά. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι είμαι ανοιχτό. Αλλά δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε από τη μια μέρα στην άλλη. Το θεσμικό όργανο της τράπεζας αυτής δεν είναι το ίδιο όπως εκείνο που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είμαστε μια χώρα. Άρα πρέπει να ληφθούν πολλοί παράγοντα υπόψη για να μην έχουμε πανεθνικοποίηση τη νομισματική πολιτική. Όλα τα μέλη πάντως του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται εκεί υπό την προσωπική τους ιδιότητα. Δεν εκπροσωπούν τις χώρες τους. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και υπάρχουν και άλλε διαστάσει που μα κάνουν να σκεφτόμαστε ότι αν το κάνουμε πρέπει να το κάνουμε με ρεαλιστικό πνεύμα χωρίς ε, φυσικά να μειώνεται σε τίποτα η διαφάνεια. Όπως και να έχει το πράγμα, το συζητάμε. Πρέπει να ξέρετε συλλογικά. Τώρα η ερώτηση που έγινε για τη διαθεσιμότητα των οριστικών νομισματικών συναλλαγών. Δεν πρόκειται για αντικατάσταση της πρόσβασης στην αγορά. Δηλαδή οι χώρες που κερδίζουν ή έχουν ήδη κερδίσει την πρόσβαση στην αγορά. Τα OMT, οι οριστικές μορφωτικές συναλλαγές, δεν αντικαθιστούν αυτή την πρόσβαση, γιατί τότε θα ήταν σαν να βρίσκονται πάρα πολύ καλά στη, στα νομισματικά, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει η συνθήκη. Τώρα για το θέμα του πώς θα υπάρχει η λογοδοσία, πώς θα είναι υπόλογος ο νέος επόπτης. Θέλουμε να είναι όσο γίνεται περισσότερο υπόλογο το νέο σχήμα όσο προχωράμε και είμαστε στα χέρια των νομοθετών εδώ. Εκείνοι πρέπει να μας πούν τι προδιαγραφές επιθυμούν. Αλλά όσον αφορά την προετοιμασία, εμείς θα συμμορφωθούμε με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Και το τελευταίο ερώτημα είναι για την προσαρμογή ή όχι. Αυτή την ερώτηση την ακούσαμε πολλές φορές. Με ρωτάτε υπάρχει πρόοδος, έχει νόημα. Γίνονται θυσίες συγκεκριμένες, πραγματικές. Υπάρχουν εδώ και καιρό που γίνονται, οπότε είναι απόλυτα φυσικό να έρθει το ερώτημα που είναι η πρόοδος. Ε, λοιπόν, σας λέω ότι έχουμε δει κάποια πρόοδο. Υπάρχουν ε, τέτοια μηνύματα, δείγματα για το εργασιακό κόστος, για την ανταγωνιστικότητα που κερδίζεται σιγά σιγά, που μειώνονται τα ελλείμματα, που αυξάνονται οι εξαγωγές. Συνεπώς υπάρχουν τέτοια δείγματα. Στην Πορτογαλία είδαμε ότι για πρώτη φορά η Πορτογαλία εξέδωσε ομόλογο στην αγορά πριν από μία εβδομάδα. Ποιος άλλος. Ιρλανδία. Α, Ιρλανδία. όπου πρώτη έκανε πρόοδο και μεγαλύτερη πρόοδο από τους υπόλοιπους. Συνεπώς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι φοβερές θυσίες που έλαβαν χώρα αποφέρουν καρπούς και πρέπει να αναγνωρίσουμε την τεράστια πρόοδο που γίνεται και όσον αφορά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και όσον αφορά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Για την Ελλάδα, ρωτάει ο κύριος Ντράγκη. Υπήρχε ερώτηση. Νόμιζα ότι υπήρχε μια ερώτηση για την Ελλάδα. Δεν υπήρχε. Πριν ήταν στον προηγούμενο γύρο, λέει ο κύριο Στράκη. Καλά, εγώ τότε θα τα έχω χάσει. Μάρτα τώρα και μετά ο Χάνς Πίτερ Μάρτιν και ο Παύλο μετά. Ευχαριστώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυτό το πρόγραμμα οριστικών νομισματικών συναλλαγών για να στηρίξει το ευρώ. Αγορές ομολόγων στις ε, δευτερογενείς ε, αγορές. Εσείς τι προσδοκίες έχετε. Πόσο θα βοηθήσει πιστεύετε αυτό το μέτρο. Δεύτερον, πώς αυτή την ρευστότητα θα την απομονώσετε. Δηλαδή, ποια θα είναι η πηγή χρηματοδότησης. Η τρίτη μου ερώτηση είχε να κάνει με το σχόλιο σας για την αρεσιμότητα, ότι επιβάλλεται στις κυβερνήσεις να αγοράζετε ομόλογα από επενδυτές. Πού θα πιέσετε ώστε οι κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με την αιρεσιμότητα. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχει μια ε, διχοτομία, δηλαδή αγοράζεται από τους επενδυτές αλλά πιέζεται τις κυβερνήσεις. Ευχαριστώ. Ο Χάντς Πίτερ Μάρτιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, ε, υπενθυμίζω το πρόβλημα των διατραπεζικών αγορών και το σύστημα του Target 2. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ανισομέρεια στο σύστημα Target 2. Και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια τεράστια μετακίνηση από τη, του κινδύνου από τις τράπεζες στις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης. Το πρώτο ερώτημα. Συμφωνείτε ότι υπάρχει αυτή η ανισομέρεια ενός, δισεκα, τρισεκατομμυρίου ευρώ και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί στην ε, Γερμανία ήδη οφείλονται ε, δισεκατομμύρια ευρώ ενώ το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας περιώσει τη συμμετοχή της Γερμανίας στα 90 δισεκατομμύρια στο σύστημα ESM ε και γιατί δεν έχει δημιουργηθεί και ένα σύστημα εξισορρόπησης όπως τις Ηνωμένε Πολιτείε ώστε να υπάρχει αυτή η... Δυστυχώς δεν μιλάω Ιταλικά κύριε Δράγη, παρακαλώ να με ακούσετε. Ένα σύστημα λοιπόν όπως αυτό που ισχύει στο αμερικανικό σύστημα και να υπάρχει μια πιο τακτική εξίσωση των υπολείπων. Γιατί στο ευρωπαϊκό σύστημα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και τρίτον, συμφωνείτε ότι λόγω αυτού του σχετικά άγνωστου συστήματος Target 2 οι χώρες οι οποίες έχουν τα μεγαλύτερα πλεονάσματα είναι εκβιάσιμες γιατί δεν τη συμφέρει η διάσπαση του συστήματος του ευρώ. Σας ζητώ να περιοριστείτε σε 1,5 λεπτό, λέει η πρόεδρος. Και έτσι να έχει 3,5 λεπτά χρόνο ο Μάριο. Αν μιλάει ο καθένας τρία λεπτά, τότε δεν θα έχει πάνω από 2 λεπτά. Παύλο. Ο Παύλο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η κρίση έχει οδηγήσει σε αναμόχλευση των παθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς υποστηρίζετε πάντα την ιδέα να μπορέσει από το 2013 να λειτουργήσει μια ένωση σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο και να μπορεί να δοθεί η απαραίτητη αρρωγή στις τράπεζες που την απαιτούν. Και εσείς έχετε υποστηρίξει αυτό το στόχο. Αλλά Υπάρχουν πολλοί από τους επικριτές σας που θεωρούν ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι προετοιμασμένη και έχει την ικανότητα ώστε μέσα σε τρεις μήνες να αναλάβει την τραπεζική εποπτεία όπως ακριβώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να ξέρω επίσης κύριε Ντράγκη αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς θα οργανώσετε αυτές τις ενέργειες. Επίση, οι νομισματικές πράξεις μαζί με τις μεταρρυθμίσεις και την δημοσιονομική εξυγίανση θεωρείται ότι είναι η λύση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κατακαιρματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αλλά το ερώτημα μου το εξή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό πέραν των οριστικών αυτών πράξεων για να ξεπεράσει τον κατακαιρματισμό των αγορών όταν δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές για να μπορέσουν να τεθούν σε λειτουργία αυτές οι οριστικές συναλλαγματικές, ε, νομισματικές συναλλαγές για μια ορισμένη χώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν αυτοί οι τρεις. Πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το σύστημα των νομισματικών συναλλαγών δεν θα υπάρχει όριο. Το μέγεθος θα είναι το κατάλληλο για να πετύχει τους στόχους της η μορφή αυτή παρέμβαση. η ρευστότητα αν θα αποστηρωθεί, όπως ακριβώς το κάνουμε και με το SNP. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια, θα έλεγα, αυθύπαρτη γέννηση ρευστότητας. Η αιρεσιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος. Είμαστε πεπισμένοι, έχουμε έτσι και αλλιώ εμπειρίες, αλλά πιστεύουμε ότι το MT χωρίς αιρεσιμότητα δεν μπορεί να υπάρξει. Για τις ανισότητες ε, και ανισορροπίες, συγγνώμη, σχετικά με τον στόχο 2. Υπάρχουν δύο λόγοι εδώ, δύο αιτίες αν θέλετε. Καταρχάς, τα διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας σε ορισμένες χώρες έχουν πλεονάσματα, άλλες χώρες έχουν έτσι και αλλιώς ελλείμματα και οι ενδοευρωπαϊκές ροές που προέρχονται από τα διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης που τρέφουν οι αποταμιευτές και οι επενδυτές στα πιστοτικά συστήματα. Έχετε λοιπόν από τη μία καταθέσεις και κεφαλαιοχικές ροές από ορισμένε χώρες προς άλλες συγκεκριμένες. Υπάρχουν όπως είπα δύο λόγοι. Ο δεύτερος λόγος είναι αυτός τον οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Εάν αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη και αν αποκαταστήσουμε εμπιστοσύνη στα πιστοτικά συστήματα της Ευρωζώνης και αναφέρθηκα στα τρία βήματα που απαιτούνται και στο πρόγραμμα αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς να εφαρμόσουμε για την απόσυρση του καθορισμένου κινδύνου, τότε πιστεύουμε ότι οι ανισορροπίες αυτές θα μειωθούν. Γιατί τα κεφάλαια δεν θα έχουν τον λόγο να μεταφερθούν από ορισμένα πιστοτικά συστήματα σε άλλα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και θα παραμένουν εκεί που είναι. Τους τελευταίους δύο-τρεις μήνες είδαμε ισροές κεφαλαίων σε κάποιες από τις λεγόμενες ευάλωτες χώρες. Και αυτό για πρώτη φορά εδώ και πάρα πάρα πάρα πολύ καιρό. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει μια ανάκτηση εμπιστοσύνης και αυτή η ανάκτηση εμπιστοσύνης επηρεάζει θετικά μειώνοντας ή σταθεροποιώντας τουλάχιστον ε, τα ποσοστά ανισοτήτων και γι' αυτό τα μέτρα τα οποία έχουμε αναγγείλει μειώνουν ακόμα περισσότερο τους κινδύνους τους οποίους εκτίθενται ορισμένες χώρες. Ο δεύτερος ε, ε, θα έλεγα λόγος αφορά ε, τα πλεονάσματα που παρουσιάζουν ορισμένες χώρες και τα διαφορά ποσοστά εμπιστοσύνης. Αν οι χώρες δεν ανακτήσουν ανταγωνιστικότητα, είναι τα πράγματα δύσκολα. Μέσα σε μια ένωση έχουμε ορισμένες χώρες που είναι μόνιμοι πιστωτές και άλλες χώρες οι οποίες ε, είναι μόνιμα δανειζόμενες χώρες. Λοιπόν, ένα τμήμα αυτής της επανεξισορρόπησης θα προέλθει από την ανάκτηση ε, ανταγωνιστικότητας και αυτός θα είναι καρπός θα έλεγα των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων και στον τομέα των αγαθών και στον τομέα των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα αναλάβει την εποπτεία μέσα σε τρεις μήνες και θα το κάνει αυτό αμέσως. Όχι, υπάρχει μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Νομίζω ότι θα χρειαστεί ένας χρόνος τουλάχιστον για να προσαρμόσουμε τις δομές που υπάρχουν για αυτό το στόχο, για αυτό το λόγο. Το σημαντικό είναι το, το κανονισμός του Συμβουλίου να τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου, σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και θα συνεργαστούμε με τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές για την αποκατάσταση του συστήματος. Πάνω κάτω θέλουμε ένα χρόνο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Για την αιρεσιμότητα πάλι. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, αλλά αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις δεν θα δουλέψουν τα OMT. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να βελτιώσει και να αποκαταστήσει τη μετάδοση των μέτρων της νομισματικής πολιτικής που λαμβάνει. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξουν αναφορές για τους λόγους της ε, ε, δυσκολίας μετάδοσης και τότε μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε, υπήρξαν πολλές ανταλλαγές ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες. Ελπίζω οι επόμενοι τρεις να είναι οι εξής. Ιντβελτ, Έπινγκ για μια ακόμη φορά. Η Μακάρτη, μια σύντομη ερώτηση. Είναι θετικό όταν βλέπει κανείς τις χώρες εκτός Ευρωζώνης στην ε, Τραπεζική Ένωση υπάρχουν δυνατότητες, αν και υπάρχουν κάποια νομικά θέματα και πρακτικά όμως θέματα πρόεδρε. Σαν παράδειγμα, οι τράπεζες στην Τσεχία ανήκουν σε ζώνες που ανήκουν στην Ευρωζώνη. Το ίδιο γίνεται και με την Εστονία με τις Σουηδικές τράπεζες. Ε, γενικά υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση ανάμεσα στην ζώνη και εκτός ζώνης. Και πρακτικά, όπως είπε και ο Σουηδός Πρωθυπουργός, τι έχουν να κερδίσουν οι χώρες εκτός ζώνης από την Τραπεζική ε, Ένωση. Θα διαβηθούν οι εγγυήσεις σας προς τα μέλη εκτός ζώνης. Ε, υπάρχουν ε, κίνδυνοι κάποιες τράπεζες να μεταφέρουν ε, τις έδρες τους στην Ευρωζώνη. Μια ολόκληρη σειρά γενικά από πρακτικά θέματα που τίθενται για τη λειτουργία των πιστοτικών ιδρυμάτων και όχι μόνο νομικά. Η Σοφία Ιντβέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ε, για την ε, Τραπεζική Ένωση, εσείς πιστεύετε ότι ένα πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων είναι βασικό χαρακτηριστικό αυτής της Ένωσης. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Γερμανία δεν θέλει να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύετε ότι τελικά μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα, αλλά πόσο ρεαλιστική είναι η προσδοκία σας και τι θα γίνει αν δεν γίνει πραγματικότητα. Θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις σας ε, για ε, τα τρία ε, γεράκια, Φιλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, ότι δηλαδή το θέμα εδώ θα πρέπει εν να παραμείνει σε εθνικό επίπεδο και δεν υπάρχει καμία σύνδεση με το ESM. Τέλος, από ό,τι φαίνεται το ΔΝΤ δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία σας κύριε Ντράγκη για τις εξελίξεις της οικονομίας. Ζητούν για εξελίξεις ολοκλήρωσης και στον τομέα των τραπεζικών αλλά ζητούν υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού για χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία μέχρι και 4% και να σταματήσουν οι πιέσεις στις μισθολογικές ρυθμίσεις. Αυτά όλα είναι αντίθετα με τη δική σας προοπτική. Πώς βλέπετε τις απόψεις του Δέλτα Ευχαριστώ. Σέπιν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σκεφτεί τι αρνητικέ ενδεχομένω επιπτώσει ε, περιορίζοντα ε, τι οριστικέ νομισματικέ συναλλαγέ μόλι αρχίσουν εφόσον ε, δεν τηρούν πια τις προϋποθέσεις οι χώρες. Δεν θα υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος. Αντιλαμβάνεστε την ερώτησή μου, Πρόεδρε. Δεύτερον, για την Πάνκια. Χτες συζητήσαμε με τον Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό, τον κύριο Αλμούνια, το θέμα και η εντύπωση μου είναι ότι η Ισπανία συγχώνευσε αυτές τις 7 περιφερειακές τράπεζες για να δημιουργήσει μια μεγάλη τράπεζα, too big to fail, πολύ μεγάλη και δεν θα, για να διατηρηθεί εν ζωή. Υπάρχουν όμως οργανισμοί όπως η ΕΛΠΑ ή ακόμη και η Real Madrid και άλλοι που έχουν τεράστια χρέη. Ποιος τελικά θα σώσει την Bankia. Αυτά τα αυτό το τοξικό ενεργητικό δεν θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, γιατί ακόμα και αν λυθεί η μπάνκια, στην ισπανική οικονομία παραμένουν τεράστια προβλήματα. Είναι σαν να ξεκολλάτε από το τοίχο ανακαθρέφτη και μετά πέσει και ο τοίχος. Για την πρώτη ερώτηση. Στις περιπτώσεις που αναφέρετε, χρειάζεται δουλειά. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ε, σήμερα πώς λειτουργεί η εποπτεία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχετε εποπτικά συμβούλια. Συμβούλια εποπτών. Και ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας θα αποτελέσει μέρος των συμβουλίων αυτών. Συνεπώς, δεν πρόκειται να υπάρξει μεγάλη αλλαγή στην δομή της εποπτείας έτσι όπως γίνεται σήμερα. Είτε πρόκειται για θηγατρικές, είτε για ξένες τράπεζες εκτός ε, Ευρωζώνης ή από τράπεζες από την Ευρωζώνη σε χώρες μη Ευρωζώνης. Υπάρχει εποπτεία μέσω των εποπτικών συμβουλίων όπου συμμετέχουν και οι αφιτριώνες χώρες και οι χώρες προέλευση των τραπεζών τώρα. Θα υπάρχει αυτός ο ενιαίος μηχανισμός και θα υπάρχει και ο διαφερόμενος επόπτης. Οπότε από καθαρά άποψη πλαισίου, το πλαίσιο υπάρχει και οι αλλαγές το ότι δηλαδή ο ενιαίος μηχανισμός θα αποτελεί μέρος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι το μόνο. Το μόνο που αλλάζει. Όσον αφορά την πρόσβαση στη ρευστότητα, η απάντηση είναι όχι. Διότι η εποπτική πολιτική έχει να κάνει με τις τράπεζες που βρίσκονται στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Τώρα για τις εγγύσεις καταθέσεων. Αυτό είναι πολύ βασικό, αλλά βασικός πυλώνας, αλλά χρειάζεται χρόνο. Όταν μιλάμε για τις εγγύσεις καταθέσεων, μιλάμε για ε, τον επιμερισμό της, ε, του τραπεζικού κινδύνου. Δηλαδή κάποιες χώρες, κάποιοι που μπορούν να σώσουν, αναλαμβάνουν, επομίζονται τον κίνδυνο ο οποίος βρίσκεται στις ε, τράπεζες στις άλλες χώρες. Πριν γίνει όμως αυτό, πρέπει θέλεις να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τι υπάρχει στις τράπεζες αυτές. Εξού και οι τρυπηλώνες που έχουν ε, να κάνουν και με τον έλεγχο και με την εξυγίανση και με την εποπτεία. Αλλά η διάφρωση θα είναι διαφορετική. Θα υπάρχει ένας ενίος μηχανισμός, ο οποίος θα κοιτάζει τι γίνεται στις τράπεζες, τι κίνδυνος υπάρχει και θα κάνει μια αξιολόγηση. Και μόνο μετά θα αποφασίζουμε για τον επιμερισμό αυτών των κινδύνων. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που γίνεται βαθμία. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τα εθνικά προγράμματα εγγύησης καταθέσεων. Όταν γίνει μεταφορά σε μια νέα οντότητα, προηγουμένως θέλουμε να ξέρουμε σε τι δεσμευόμαστε. το τι έχουμε κληρονομήσει από παλιά. Ε, τι είναι αυτό που έχουμε κληρονομήσει από παλιά και τι δεν είναι, πώς γίνεται αυτή η διάκριση. Αυτή η διάκριση εκπλήσει μερικούς και πρέπει να διευκρινιστεί, αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να διευκρινιστεί πράγματι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά τώρα ανάμεσα στις προβλέψεις για την ανάπτυξη του Διεθνούς Ομοσπονδιακού Ταμείου και των δικών μας βγαίνουμε από το δεύτερο τρίμηνο με μια πολύ αδύναμη δραστηριότητα. Το επόμενο μάλλον το ίδιο θα έχουμε, οπότε ε, δεν θέλω να φανώ υπερβολικά αισιόδοξο όσον αφορά την ανάπτυξη. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, μην ξεχνάμε ότι η εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να κρατάει τον πληθωρισμό για την Ευρωζώνη κάτω ή τέλο πάντων κοντά στο 2% για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αυτή είναι η εντολή. Τώρα, τι γίνεται με τον πληθωρισμό σε διάφορες ε, χώρες, αποτελεί αυτό ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εφόσον έχει να κάνει με την εξέλιξη των τιμών σε κάποιους τομείς. Αυτό μέσω μακροπροβλητικής εποπτείας πρέπει να αντιμετωπιστεί αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής γίνεται σε εθνικό επίπεδο, με κεντρική βοήθεια από εμά. Δηλαδή, καταρχήν η εντολή μας είναι για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Η επόμενη ερώτηση για τις οριστικές νομισματικές συναλλαγές, τα OMTs. Δεν θυμάμαι όμως τι ακριβώς με ρωτήσατε. Η ερώτηση ήταν η εξής. Άπαξ και τα έχετε προσφέρει αυτά, θα αναγκαστείτε ίσως μερικές φορές να τα κόψετε. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος, θα μπορέσετε να τα κόψετε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αντιμετωπιστεί από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και θα σας διαβάσω την ανακοίνωση που έκανα εγώ όταν είχαμε τελευταία συνέντευξη τύπου. Λέμε ότι αυτές οι συναλλαγές δεν θα λάβουν χώρα εφόσον υπάρχει αναθεώρηση κάποιου προγράμματος εξυγένσης και θα ολοκληρώνεται μετά την περίοδο αναθεώρησης εφόσον έχει διασφαλιστεί ολοκλήρωση του προγράμματος. Δηλαδή δεν θέλετε να έχετε τέτοιες συναλλαγές όταν υπάρχει αναθεώρηση επιτόπου, γιατί γίνονται πολλές διαπραγματεύσεις και πολλοί παράγοντες που μπορεί να αλλάξουν στο μεταξύ. Αλλά εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική, τότε θα ξαναρχίζουν. Για την μπάνκια τώρα και το ρευστό. Η ερώτησή σας έχει να κάνει με τους ε, κινδύνους οι οποίοι έχουν συσσωρευτεί. Ξέρετε ότι η Ισπανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνουν διαπραγματεύσεις και συζητήσεις για τη δημιουργία μιας ε, επιχείρησης όπου κάποιο ενεργητικό κάποιων ε, τραπεζών, μεταξύ άλλων και της Μπάνκια, θα μεταφερθούν εκεί. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό εγώ τώρα να συζητήσω ή να σχολιάσω για διαπραγματεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ο επόμενος γύρος, ο Μάριο Μάουρο, ο Ούντο Μπούλμαν και η Αστρίδ Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. επανέρχομαι στο θέμα της αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων γενικότερα. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις που δώσατε ήδη, αλλά να θέσω μια άμεση, θα έλεγα, ερώτηση. Νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο ότι το θέμα της αιρεσιμότητας εμπεριέχει μια κάποια μεταφορά κυριαρχίας σε εθελοντική βάση κάτι το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση όχι τόσο το νομικό κομμάτι της ενέργειας, αλλά το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου και της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Δεν θα ήταν ε, καλό οι χώρες μέλος να νομιμοποιήσουν αυτού του τύπου τις αποφάσεις και διαδικασίες με μία αλλαγή στις συνθήκες και όχι να λέγουν ότι απλά μέσω της ερεσιμότητας θα έχουμε μια συνεχή διακύμανση στην εφαρμογή των συνθήκων, μιας και ασχολούμαστε με θέματα τα οποία δεν είναι θα έλεγα αυτόματα κάτι το οποίο ανάγκη στην ευρωπαϊκή κυριαρχία. Και δεύτερον, τι γίνεται με τις κεντρικές δημόσιες επενδυτικές τράπεζες όπως οι τράπεζες παρακαταθήκων και δανείων, οι οποίες πολλές φορές λειτουργούν με δικό τους ξεχωριστό κομμάτι στον προϋπολογισμό. Ο Μπούλμαν. Και εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να φορέσετε τα ακουστικά σας και να με ακούσετε γιατί θα μιλήσω γερμανικά και Πρόεδρε παρακαλώ να αρχίσει από τώρα η χρονομέτρηση της ομιλίας μου. Κύριε Πρόεδρε, εγώ μπορώ να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μάουρο με το θέμα της ερεσιμότητος. Αν τελικά αυτό το οποίο θα προκύψει είναι μια νέα μορφή διακυβέρνησης στον οικονομικό χώρο, τότε φυσικά εσείς ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορείτε να διεκδικήσετε ένα σημαντικό τμήμα αυτής της διακυβέρνησης και εσείς έχετε λόγο να σας επενέσουμε για τις προηγούμενες δράσεις σας και έχετε πράγματι κερδίσει μια θέση για τα θέματα αυτά. Αλλά όλα αυτά τα ζητήματα, το σύστημα σταθεροποίησης, το θέμα της ε, αιρεσιμότητας, όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε. Είναι καλό για όλους μας να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό σχήμα Διακυβέρνηση το οποίο θα εμπεριέχει και την ερεσιμότητα. Υπάρχει όμως ένα κέριο πρόβλημα και εσείς ως εκπρόσωπος του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είστε κομμάτι αυτού του προβλήματος. Η ερεσιμότητα είναι μια πολιτική διατύπωση κατά κάποιο τρόπο, μια ε, επιβολή στον οικονομικό στίβο που μπορεί να είναι και λανθασμένη όταν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κάνει λάθη, μπορεί να χάσει τις επόμενες εκλογές. Τα κοινοβούλια επίσης μπορούν σε μια επανεκλογή να χάσουν τη θέση τους οι βουλευτές. Αλλά η Τρόικα είναι ένας μη εκλεγμένος φορέας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει λύσεις στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Μα εδώ δεν έχουμε ένα κράτος όπου είναι οι σοφοί οι οποίοι διοικούν την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι φορείς για απάντηση είναι οι κυβερνήσει και τα κοινοβούλια. Αυτή είναι δημοκρατικά υπεύθυνη. Γιατί λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχει αυτή η κατάσταση και πρέπει η Επιτροπή μας να έχει και αυτή κάποιο ρόλο για να εξετάσει το πώς επιβάλλεται η αιρεσιμότητα, πώς γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στα προγράμματα αυτά και αυτό προς το συμφέρον των πολιτών των χωρών που βρισκόνται επιτήρηση. Αν θέλουμε να έχουμε μια υπερεθνική εξουσία πρέπει να υπάρχει έλεγχος κοινοβουλευτικός από ένα υπερεθνικό κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Ντράγκη, η εκστρατεία για μια γυναικεία παρουσία στο διοικητικό σας συμβούλιο η οποία αποστέρισε από τον κύριο Μέρς για κάποιους μήνες τη θέση του παρά τις ικανότητες του που είναι αδιαφυσβήτητες είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί και ο μύθος της γυναίκας η οποία έχει όλες τις αρετές ενώπιον ανδρών που είναι γεμάτοι ψεγάδια. Θυμάμαι αυτά τα οποία έλεγε η κυρία ε, Ρέντινγκ που έλεγε ότι αν ήταν γυναίκες οι οποίες είχαν την εξουσία στους Lehman Brothers, οι Lehman, ήταν οι αδερφές Lehman και όχι οι αδερφοί Λέμαν δεν θα είχαν υπάρξει τόσα πολλά προβλήματα. Και επανέρχομαι στο θέμα αυτό της κρίσης του 2008 είναι δύο γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα κέντρα των σκανδάλων των ε, Lehman Brothers και της Goldman Sachs που τις ξέρετε και καλύτερα από μένα τον, την ίδια. Εγώ θα μπορούσα να σας περιγράψω τι έχουν κάνει, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά σας ζητώ να διαβάσετε αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που έχει τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί. Για να σας πω ότι θα έπρεπε και εδώ να δείτε τα γεγονότα προτού κάνουμε γενικεύσεις. Και δεν μπορούμε να λέμε αερολογίες. Για μένα είναι σημαντικό. Ξέρετε ότι εγώ από την αρχή της πολιτικής μου καριέρας, το 1963 μάλιστα, αγωνίζομαι για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βασιζόμαστε πάντα επί πραγματικών γεγονότων γιατί ένας ευγενής αγώνας πρέπει να βασίζεται πάντα στην αλήθεια και όχι σε μυθολογίες. Και θέλω να σας θέσω λοιπόν ένα ερωτηματάκι κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για την αρχή της αποκέντρωσης η οποία θα εφαρμοστεί στα πλαίσια του μηχανισμού εποπτείας, του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας. Πώς η Κεντρική Τράπεζα λοιπόν μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι εθνικές αρχές εργάζονται εποφελώς μέσα στο σύστημα αυτό και δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά εθνικά συμφέροντα στις χώρες όπου εργάζονται. Γιατί αν κατανοώ καλά τα πράγματα, θα πρέπει να υπάρξει κάποιος διάλογος, ο οποίος να είναι ιδιαίτερα έντονος μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Εποπτικών Αρχών, αλλά γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι αυτή που σε τελική ανάλυση θα έχει την ευθύνη και θα πρέπει να έχει τους απαραίτητους πόρους για να εφαρμόσει αυτήν την τελική της ευθύνη. Ωραία. Έχετε το λόγο κύριε Δράγη. Για τα πρώτα δύο ερωτήματα. νομίζω ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία τα ερωτήματα αυτά. Έχουμε επιχειρηματολογήσει κάθε επανάληψη, κατά συρροή, ότι πρέπει να υπάρξει μια από άσκηση της κυριαρχικότητας σε ένα υπερεθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό, τον φορολογικό και τώρα όλο και περισσότερο στον τομέα των οικονομικών διαρθρωτικών αλλαγών. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μας πείσετε γιατί είμαστε απόλυτα πεπισμένοι για την ανάγκη αυτή. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε μπορεί να επιτευχθεί στο χώρο αυτό θα είναι μια μείζον βελτίωση για την διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι πάντα προς την, δική σας, από τη δική σας μεριά για τα θέματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά που κάνετε για τις οριστικές νομισματικές πράξεις και την ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού. Θα σας πω και πάλι ότι δεν είμαστε εμείς που επιβάλλουμε τις προϋποθέσεις. Θέλουμε απλώς να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμά μας είναι αποτελεσματικό, παραμένει μέσα στην εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν υποκαθιστά δράσεις κυβερνήσεων ή αδράνεια κυβερνήσεων αν θέλετε. Από αυτή την ε, οπτική γωνία λοιπόν η ερεσιμότητα η οποία συνοδεύει τις οριστικές νομισματικές συναλλαγές έχει θεμελιώδη χαρακτήρα. Ξέρουμε ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα λειτουργήσουν. Το ξέρουμε από την πείρα. Και απλά από μια θεωρητική ανάλυση μπορούμε να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα ότι οι, οι νομισματικές συναλλαγές δεν θα ωφελήσουν χωρί μια αρεσιμότητα, γιατί θα καταστρέψουν τα κίνητρα, όπως έγινε πέρσι σε συγκεκριμένε θα καταστρέψουν τα κίνητρα για κάποιες κυβερνήσει να δράσουν και να εφαρμόσουν τις απαραίτητε μεταρρυθμίσει. Αλλά ατενίζοντας το μέλλον, πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να έχουμε ένα υπερεθνικό μηχανισμό από κοινού διαμοιρασμού της κυριαρχικότητας στους τομείς αυτούς, τόσο το καλύτερο. Οι χώρες μας είναι πια τόσο αλληλένδετες και τόσο διασυνδεδεμένες, δεν μπορούν πια να παίρνουν οικονομικές αποφάσεις οι οποίες θα έχουν αρνητικά αποτελέσματα σε άλλες χώρες που θα είναι κυρίως αρνητικού χαρακτήρα. Πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν την καθαρά εθνική οπτική γωνία όταν σχεδιάσουμε και όταν εφαρμόζουμε οικονομικές πολιτικές. Για το τελευταίο ερώτημα, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα τι εννοούσατε, αν μπορώ να σας ζητήσω, κυρία Λούλινγκ, να επαναλάβετε. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Είχα ένα συγκεκριμένο ερώτημα, λέει η κυρία Λούλινγκ, ακόμα χωρίς μικρόφωνο. Ανα... Αναφέρθηκα στο μύθο των των γυναικών και των ψεγαδιασμένων ανδρών και έκανε και κάποια αναφορά στο, στην προέλευση ορισμένων από την Goldman Sachs. Λοιπόν, σας το ξαναλέω. Γιατί θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερο για την αρχή της αποκέντρωσης που θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα στα πλαίσια του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας. Πώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι οι εθνικές αρχές εποπτείες εργάζονται πράγματι προς όφελος του συστήματος και δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα εθνικά συμφέροντα στις χώρες όπου λειτουργούν. Και ήθελα να σας πω ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένας ιδιαίτερα στενός και έντονος διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Αρχών Εποπτείας γνωρίζοντας πάντα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι ο τελικός υπεύθυνο για οποιαδήποτε ενέργεια ελέγχου και επομένως θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα μέσα για να ασκήσει αυτή την ευθύνη. Καπίτο, ε, κουέστο! Σας ζητώ. Συγγνώμη που... Που δεν κατάλαβα στην αρχή το ερώτημα σα όντω. είναι κάτι που πρέπει να φροντίσουμε και θα το φροντίσουμε μέσω της πίεσης ομολόγων peer pressure. Βλέπετε όταν θα λειτουργεί πλήρως το σύστημα αυτό, τότε θα οδηγήσει σε πολύ ανοιχτή ανταλλαγή ανάμεσα στους επόπτες όσον αφορά για την καλή κατάσταση των οργανισμών των οποίων είναι επικεφαλής. Οπότε αυτή η πίεση ομολόγων, οι ανταλλαγές απόψεων, οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από κοινό, δεν υπάρχει καμιά εμφιβολία ότι θα ξεπεράσουν την τάση αυτή που λέτε που θα είναι δεχομένω ε, που θα ε, βοηθήσουν να υπάρξει μια σωστή απόφαση. Πιστεύω ότι θα γίνει με πολύ επικοδομητικό τρόπο και θα καταφέρουμε όντως να φτιάξουμε πολύ καλά αυτόν τον ε, ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Σίγουρα θα είναι μια θετική έκπληξη. Ευχαριστώ. Καλώς, λέει η Πρόεδρος. Μπορούμε και τους υπόλοιπους ε, ομιλητής να τους ε, ακούσουμε. Πείτε Σίμων, Ιωγοφέο και Λία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Δύο θέματα. Ναι. Για το θέμα της εποπτείας υπάρχει το ζήτημα ε, της σημασίας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για τα άλλα κράτη-μέλη που είναι εκτός του, της ζώνης του ευρώ δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποια λύση. Το ερώτημα μου τώρα είναι το εξής ποιος είναι ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στο γενικό σύστημα, αυτό έχει φανεί από την ε, απόφασή της να προβεί σε αγορές ομολόγων απεριόριστα. Και έτσι κατάφερε αυτό το οποίο δεν είχαν καταφέρει οι κυβερνήσει στην αγορά τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή να μειώσουν τα επιτόκια. Τώρα, αν εσείς αναλάβετε στον εποπτικό μηχανισμό και συνεργάζεστε με εθνικές αρχές οι οποίες λειτουργούν αλλού καλά, αλλού καλά και αλλού όχι καλά. Μήπως ο μηχανισμός αυτός θα υπόκειται και αυτό στο μέλλον και μήπως θα υπάρξουν και στο μέλλον νέε κρίσεις, ίσως λιγότερες από ό,τι τώρα λόγω του καλύτερου μηχανισμού. Ε, γιατί τώρα οι άνθρωποι που θα αναλάβουν τις αναδιαθρώσεις των τραπεζών είναι αυτοί οι οποίοι ήδη ασκούν τώρα εξουσίες οι οποίες έχουν αποτύχει στα κράτη-μέλη πολλές φορές. Μήπως φοβόσαστε ότι στο μέλλον θα υπάρξει έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών ε, στον φορέα αυτό, γιατί ακριβώς θα στελεχώνεται με άτομα τα οποία έχουν κάνει λάθος στο παρελθόν, τα οποία έχουν χάσει χρήματα κτλ. κύριος Φέιου. Ευχαριστώ Σιάρουν και τον ε, κύριο Ντράγκη. Θέλω να σας ε, ευχαριστήσω για τις απαντήσεις σας. Προηγουμένως αναφέρθηκε στο ερώτημα σε σχέση με την κατάσταση της Πορτογαλίας. Λέτε ότι υπήρξε έκδοση χρέου η οποία ήταν επιτυχής και επίσης η πέμπτη αξιολόγηση της Τρόικα ήταν θετική και δόθηκε και μία ακόμα ε, δόση χρηματοδότηση στην Πορτογαλία. Και με όλα αυτά, ελπίζετε ότι η Πορτογαλία θα μπορέσει να ξαναγυρίσει στις αγορές του Σεπτέμβριου 2013 όπως προβλεπόταν. Είναι πράγματι η Πορτογαλία στο σωστό δρόμο για να το πετύχει αυτό. Δεύτερον, ερώτημα. Έχουν ακουστεί κάποιες επικρίσεις για το μοντέλο προσαρμογής που έχει επιβάλει η Τρόικα. Περισσότερη ύφεση, περισσότερη ανεργία, μία συρρήκνωση της εσωτερικής ζήτησης καταστάσεις ρήξης σε πολλές χώρες. Μήπως υπάρχει κίνδυνος όταν οι χώρες τελειώσουν αυτή τη διαδικασία προσαρμογής δεν θα μπορέσουν να ανακάμψουν. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημα. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν στους πολίτες των κρατών μελών που υπόκειται σε τόσο μεγάλες θυσίες ότι θα μπορέσουν στη συνέχεια να βρουν το ρυθμό της ανάπτυξης. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αγοράσει εκ νέου ελληνικό χρέος. Το έκανε με πλεονεκτικό, θα έλεγα, ε, επιτόκιο και έτσι όταν λήξουν οι τίτλοι αυτοί, από ό,τι φαίνεται θα δημιουργηθεί μια υπεραξία 11 δις να προσθέσουμε και στα πλαίσια του S&P ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει την απόδοση των επιτοκίων της κατά 3,5 περίπου δις. Λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξή. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεσμεύεται από τους κανονισμούς λειτουργίας της, αλλά δεν είναι μια απλή επιχειρηματική τράπεζα, δεν είναι μια εμπορική τράπεζα, ε, και εξαιρέθηκε από την αναδιάφραση του ελληνικού χρέους τον Φεβρουάριο. Λοιπόν, έχετε σαν στόχο την δημιουργία τέτοιου ύψους κερδών. Μήπως τα χρήματα αυτά θα μπορούσατε να τα ξαναδώσετε στην πραγματική οικονομία. Μια πραγματική οικονομία η οποία υφίσταται μεταρρυθμίσεις, των οποίων οι επιπτώσεις, όπως βλέπουμε στο θέμα της ανάπτυξης, είναι θα έλεγα σε πολύ κακή φάση. Λοιπόν, τι θα κάνει αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αν αυξηθούν τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται η Ισπανία και αν η Ισπανία εξακολουθώντας να φοβάται να στιγματιστεί δεν προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Τι θα κάνει η τράπεζά σας. On, on the first question, um, Για την πρώτη σας ερώτηση. Νομίζω ότι το θέμα της εποπτείας εδώ είναι σημαντικό. Έτσι θα αποτρέψουμε δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστα λάθη. Πολλές φορές οι τράπεζες όμως ε, αποτυγχάνουν, ανεξαρτήτως της ποιότητας της επίβλεψης, της εποπτείας. Γι' αυτό λοιπόν να υπάρχει μία αρχή θα έλεγα επίλυσης προβλημάτων είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι θα δώσουμε την δυνατότητα στις κυβερνήσεις την απόλυτη ελευθερία να αφήσουν τα ιδρύματα που αποτυγχάνουν, που θα πτωχεύσουν δηλαδή, να το κάνουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο χρήμα και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στους μηχανισμούς πληρωμής που είδαμε στην περίπτωση της Lehman Brothers ή και σε περιπτώσεις επίσης μικρότερων τραπεζών. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικότατος πυλώνας ε, της, ε, ε, ε, της ένωσης αυτής της τραπεζικής που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Να μην ξεχάσουμε τι συνέβη στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες κλείσαν περίπου τα τελευταία χρόνια 200 τράπεζες. Και δεν υπήρξαν τελικά πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο σύνολο του συστήματος πληρωμών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το σκέλος της ε, ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Για την Πορτογαλία. Να πω ότι το πρόγραμμα σταθεροποίησης πηγαίνει γρηγορότερα από όσο περιμέναμε. Η οικονομία αποκαθιστά την ισορροπία της από μια οικονομία που ήταν εσωστρεφής σε μια οικονομία ε, εξαγωγική. Βλέπουμε βελτιώσεις ε, στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, μείωση του κόστους εργασίας, μείωση του ελλείμματος. Όλα αυτά είναι μηνύματα πρόοδου. Το έλλειμμα από ό,τι φαίνεται θα κατέβει κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2014 στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Η στάση της τράπεζάς μας σε σχέση με την Πορτογαλία είναι να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη μορφή πρόοδου και να ζητά την ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων Το καλό λοιπόν είναι ότι η Πορτογαλία εξέδωσε ένα ομόλογο την προηγούμενη εβδομάδα, τριετές, αν άκουσα καλά τριετές, και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση βρίσκεται σε καλή θέση να προβλέψει την επανεισδοχή της στις αγορές όπως είχε προβλεφθεί στα πλαίσια των υπαρχουσών προβλέψεων. Αυτό είναι καλό και θετικό. Και η Ιρλανδία είναι ένα παράδειγμα στο οποίο οι θυσίες θα έλεγα που γίνονται δεν είναι αυτός σκοπός. Όπως σας είπα και εγώ και όπως μου θυμήσατε ε, τις λέξεις που χρησιμοποίησα, οι θυσίες αυτές έχουν οδηγήσει πολλές χώρες τα μισά του δρόμου. Εξακολουθούν βέβαια να αντιμετωπίσουν ανέμους αντίθετους ισχυρούς, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η άλλη πλευρά του ποταμού τον οποίο διασχίζουμε. Και νομίζω ότι ε, βλέπουμε πού πάμε τώρα με βήματα προόδου και στον τομέα της ε, ε, ευρωδιακυβέρνησης. Βλέπουμε τι ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε ε, σε 5-10 χρόνια. Θυμάστε ότι από την τελευταία συζήτηση εδώ και 5-6 μήνες τα πράγματα ήταν λιγότερο καλά. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να είναι κανείς υπεραισιόδοξος, αλλά μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο ότι σημειώσαμε πρόοδο τους τελευταίους 5-6 μήνες και σε εθνικό επίπεδο με μονομένες χώρες και σε επίπεδο ευρωδιακυβέρνησης, ευρωπαϊκό επίπεδο και οι κυβερνήσεις επιμέρους τα πήγαν καλά και στα πλαίσια της προσπάθειας σχεδιασμού ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου που στοχεύει στην μελλοντική μακροπρόθεσμη λειτουργία. Τώρα, για τα κέρδη από το S&P, τα κέρδη τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, μοιράζονται στις, στα τμήματα που ανήκουν και που είναι μέλη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Διανέμονται ανάλογα με την κεφαλαιοχική τους κλίδα. Και ε, τώρα από εκεί και πέρα τι ρυθμίσεις εθνικές έχουν τα κράτη-μέλη, τα κέρδη αυτά μεταφέρονται στις κυβερνήσεις και στον υπολογισμό της χώρας και οι κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν με τα κέρδη αυτά. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις οι κυβερνήσεις δέχονται την ιδέα ότι τα κέρδη αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στη χρηματοδότηση δημοσιονομικών προγραμμάτων εξυγίανσης στις διάφορες χώρες. Σε άλλες περιπτώσεις απλά μπαίνουν ως έχουν στον εθνικό προϋπολογισμό. Δεν θέλω τώρα να κάνω προβλέψεις για το τι θα συμβεί. Αλλά τα OMT στα οποία έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε θα είναι θα έλεγα ένας καλός τρόπος για την χρήση των ευρωπαϊκών οικονομικών δυνατοτήτων. Είπαμε, δεν υπάρχει όριος προς τη χρήση αυτών των τελικών οριστικών νομισματικών συναλλαγών, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις. Και έτσι θα βοηθήσουμε έτσι ώστε να απομακρυθούν οι κίνδυνοι και να λειτουργήσουν σωστά τα συστήματα αυτά παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις που πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ευχαριστούμε. Ο Χόκμαρ και μετά και εγώ ίσως μία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, δύο πράγματα θέλω να σα ζητήσω να σχολιάσετε. Πρώτον, σε πολλέ συζητήσει που έχουμε για την Τραπεζική Ένωση, ακούγονται προτάσεις ότι κάπου, φαντάζομαι, δεν θα μπορούμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες που υιοθετούμε σήμερα. Για παράδειγμα, η για 60% όπου μιλάμε για, την, ε, για το καταμερισμό του κινδύνου. Από τη μια μεριά λοιπόν από τη μια μεριά λοιπόν προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό και από την άλλη μεριά να φτιάξουμε έναν οργανισμό ο οποίος να λύσει τα προβλήματα εκείνα που θα δημιουργηθούν εφόσον πολλές χώρες δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στους κανόνες μας. Μα δεν υπονομεύουμε έτσι αυτά που εμείς κάνουμε. Μήπως έχουμε φτιάξει υπερβολικά πολλά συμβούλια τελικά και έτσι πλήττεται η αξιοπιστία των οργάνων που ήδη έχουμε φτιάξει. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο είναι κάτι σε σχέση με αυτά που συζητήσαμε εδώ. Το μακροοικονομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές χώρες μέλη και μεγάλες οικονομίες αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι το 2020 αν κρατήσουμε το επίπεδο του 60%. Αυτό σημαίνει ότι μακροοικονομικά μιλώντας θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος. Και Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τραπεζική νομοθεσία, τις κεφαλαϊκές ε, απαιτήσεις, πράγματα τα οποία σίγουρα είναι πολύ λογικά, αλλά όλα αυτά τα υιοθετούμε συγχρόνως. Και έτσι φοβάμαι ότι η δυσκολία επιστοτική θα είναι διπλή. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, για να υπάρχει μια ισορροπία. Η Πρόεδρος. Εντάξει. Η Αρλίν σας έχει ρωτήσει ήδη. για το γεγονός ότι μπορούν να υπάρχουν μικτές ομάδες με χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Σουηδίας. Επίσης όταν μιλούσατε για την δίκες Είπατε ότι οι, ζων, οι τράπεζες της Ευρωζώνης είναι τελείως διαφορετικές από αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. γιατί έχουν ε, οι τελευταίες χώρες πολλές διεθνείς τράπεζες. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πώς εμείς θα κρατήσουμε από κοινού την ε, ενιαία αγορά με ένα, συνό, με σύνολο κανόνων που να λειτουργεί σε όλη τη ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε μια ευρύτερη περιοχή Ευρωζώνης. Ενώ λέτε ότι υπάρχουν μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι οι οποίοι είναι έξω από το πλαίσιο αυτό και μπορούν να υπάρξουν διακινήσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και αυτό θέλουμε να αποτρέψουμε. Θέλουμε να κρατήσουμε την κοινή αγορά ενιαία. Νομίζω ότι η πρόταση του κοινού εγκολπίου είναι ε, μια καλή πρόταση για να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Και έτσι μπαίνετε σε ένα πιο ε, εξελιγμένο επίπεδο μεθοδολογίας αντιμετώπισης κινδύνων που αναφέρεται στην ε, πρόταση της Κομισιόν και που ξέρω και ο η Ανδρέα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και που ήδη έχω αναφερθεί στο θέμα αυτό των ασφαλιστικών τραπεζών και κάτι ακόμα το οποίο με ενοχλεί και ενοχλεί όλους μας που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, βέβαια είναι πάρα πολλά αυτά που μας απασχολούν για την Τραπεζική Ένωση, είναι ότι και τα τρία τμήματα της Τραπεζικής Ένωσης δεν θα συγκροτηθούν συγχρόνως. Υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις για μια κοινή εποπτεία άμα δεν έχουμε κοινά αναχώματα είναι δύσκολο να έχουμε ένα νομοθέτημα, λες και η επόμενη φάση θα έρθει νομοτελειακά όταν δεν ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει κατά ανάγκη κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρξει ένα ανάχωμα θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο. Αν δεν καταφέρουμε να έχουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία, δεν μπορούμε να έχουμε την εντύπωση ότι θα είναι σίγουρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να νομοθετούμε θεωρώντας ότι κάτι θα έρθει στη συνέχεια. Αυτό από νομική άποψη δεν ευσταθεί και είναι λιγάκι σαν την μίγα στο γάλα αυτή η κατάσταση που βλέπουμε. Σας ευχαριστώ λέει κύριος Δράκη για το πρώτο ερώτημά σας. Αν κατανοώ καλά, η κύρια ανησυχία σας από ό,τι καταλαβαίνω είναι το πιο δύσκολο τμήμα της ε, η οικονομικής μας δράσης, δηλαδή η θέση από κοινού του, των κινδύνων. Για μένα όμως είναι σημαντικό αυτό, είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συγχρόνως. Για πολλούς είναι απαραίτητο να γίνει αυτό μονάχα στο τέλος των ενεργειών για την πρόοδο που έχουν γίνει. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μια συμβαστική λύση για τα θέματα αυτά αλλά όπως και στην περίπτωση του τραπεζικού συστήματος, όπου θέλαμε να έχουμε το κοινό σύστημα εγγυήσεων, η θέση από κοινού βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι όλα τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι οι οικονομικές πολιτικές είναι στοιχείο κοινού συμφέροντος. Όλα αυτά βασίζονται στην κοινή κυριαρχικότητα, ιδίως στον τομέα το χρηματοπιστωτικό, το δημοσιονομικό μάλλον και τον ε, φορολογικό. Αλλά αυτό αφορά και τις διαρθρωτικές αλλαγές. Είναι σαφές ότι θα πρέπει οι χώρες μέλη να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Και αυτό πρέπει να γίνει τμήμα του κοινού συμφώνου, επί τη βάση του οποίου θα οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη. Όλα τα προβλήματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με, το, με την κοινή διαχείριση των κινδύνων βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο αυτό. Είναι μια διαδικασία που θα χρειαστεί χρόνο, θα χρειαστεί αποφασιστικότητα, κυρίως όμως θα απαιτήσει πολιτική θέληση για να υπάρξει από κοινού θέση της κυριαρχικότητας. Και το, και το ανέφερα αυτό στο παρελθόν, θα πρέπει να γίνει αυτή η δημιουργία κοινή κυριαρχικότητα σε υπερεθνικό επίπεδο. Και το ερώτημά σα επίση έχει σωστή επιχειρηματολογία. Έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν προσπαθώντας να επιβάλλουμε κάποιες μορφές ρύθμισης ή κάποιες ειδικέ εποπτικές αξιολογήσεις οι οποίες κατέληξαν να είναι υπερκυκλικές και να επιδεινώνουν την κατάσταση. Το συζητήσαμε αυτό και στο παρελθόν. Πολλά πράγματα είναι στο χαρτί θετικά. Όταν εφαρμόζονται όμως την πράξη σε εφαρμογή πολιτικών <clears throat> θα πρέπει να εφαρμοστούν με το σωστό τρόπο και με τη σωστή χρονική σειρά. Κάτι το οποίο είναι σωστό αλλά γίνεται σε λανθασμένη χρονική στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες. Το ξέρετε αυτό γιατί έχουμε ανταλλάξει απόψη για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό πάντα τονίζω την ανάγκη να ακολουθήσουμε τη σωστή σειρά ενεργειών σχεδιάζουμε ρυθμιστικές πρόνοιες, θα πρέπει να ξέρουμε τι προϋποθέτουν αυτές οι ρυθμίσεις, τι πρέπει να υπάρχει ήδη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη βάση. Και γι' αυτό εγώ συμμερίζομαι απόλυτα και να κάνω τώρα μια σύντομη διευκρίνηση, λέει ο κ. Το πρώτο ερώτημά μου αφορούσε το γεγονός ότι πολλές από τις συζητήσεις για την θέση από κοινού του χρέους αφορούσαν το τμήμα του χρέους που ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ. Συγχρόνως, όμως το Σύμφωνο Σταθερότητας λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει χρέος που να ξεπερνάει το 60%. Και το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας τονίζει ότι το 60% πρέπει να είναι το ανώτατο όρο το, το ανώτατο όριο για το χρέος, αυτό δημιουργεί κάποια αντίφαση. Δεν θέλω να συζητήσω συγκεκριμένες λύσεις για την θέση από κοινού του χρέους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες οι οποίες έχουν προταθεί. Νομίζω ότι όλες συμμερίζονται τα προβλήματα τα οποία ανέφερα προηγουμένως. <clears throat> το ποια θα είναι η τελική απάντηση, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και να μας προβληματίσει. Και θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις αντιφάσεις μεταξύ διαφορετικών απόψεων για την ενιαία αγορά. Έχετε δίκιο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν δημιουργούμε ένα σύστημα όπου έχουμε ρυθμιστικό αρμπιτράζ ή μετακίνηση από τον ένα ρυθμιστή στον άλλο, κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει την κοινή ε, αγορά. Το να έχουμε ένα κοινό εγχειρίδιο, ένα κοινό εγκόλπιο για όλους τους ρυθμιστές, αυτό είναι όλους τους επόπτες είναι πολύ σημαντικό και όλοι πρέπει να εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό, αυτή αυτός ο νέος ενιαίος εποπτικός μηχανισμός από μόνος του δεν πρόκειται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην ενιαία αγορά από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν. Οι πραγματικότητες στον τραπεζικό τομέα είναι διαφορετικές που πρέπει να τύχουν εποπτείες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια μορφή ρύθμισης ή ένα κοινό εγχειρίδιο που θα μπορέσει να επιτύχει τα αποτελέσματα που θέλουμε, ενώ συγχρόνως σέβεται τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα που έχουμε σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η πρόταση κοινού εγχειριδίου για μένα είναι πάρα πολύ θετική και επομένως αξίζει της υποστήριξής μας. για το νομοθετικό, για το θέμα της νομοθεσίας. Από νομοθετική έποψη θα ήταν πολύ καλύτερα αν θα μπορούσε κανείς να περάσει νομοθετικά και τους τρεις πυλώνες από κοινού. Και το να κινηθούμε βήμα με βήμα είναι το πιο ρεαλιστικό, αλλά σίγουρα δυσκολεύει και τη δική σας ζωή και τη ζωή άλλων νομοθετικών οργάνων. Και σίγουρα η διαδικασία θα είναι πιο βραδία. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και η κυρία Μπάουλς. Βέβαια με την καθυστέρηση αυτή είναι δύσκολο να πετύχουμε το στόχο της 1ης Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Είναι μια χαρά για όλους μας να είστε εδώ. Και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε διάφορες ενεργητικές προσπάθειες για πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και η ισότητα των φύλων.